Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα περάσουμε στο σημείο 11 και 12 με θέμα τη μελέτη για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο. Και το σημείο 12, με ποιου τρόπου μπορεί και η γεωργική πολιτική να συμβάλλει στη δημιουργία απασχόληση στην Ήπεθρο. Έχουμε τον κύριο Μάουρο Βιγκάνη από το Πανεπιστήμιο του Σάιρ και τον κύριο Μπέρντ Σου από το Αυστριακό Ινστιτούτο Χωροταξίας. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές ζώνες, στην Ήπεθρο γενικώ. Μετά την παρουσίαση της μελέτης, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντουριουέ, τον αντιπρόεδρό μας, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Θα γίνει κοινή συζήτηση για τα δύο θέματα, γιατί είναι πραγματικά αλληλέντατα. Απλώς εξετάζουν το ίδιο ζήτημα υπό διαφορετικές σκοπιές. Ο κύριος Αντουριέ ε, θα το δει υπό το πρίσμα της πολιτικής και οι εμπειρογνώμονές μας ε, το, από την επιστημονική σκοπιά περισσότερο. Σας ε, έχουμε στείλει και υλικό ηλεκτρονικά. Τη σχετική μελέτη δηλαδή σε PDF. Δεν είναι ακόμη έτοιμα τα έγγραφα. Θα δώσω το λόγο στους δύο εμπειρογνωμονές μας, τον κύριο Μπεν Σου και τον κύριο Μάουρο Βιγκάνη, από 10 λεπτά ο καθένας. Σας ζητώ συγγνώμη που έχουμε μόνο 20 λεπτά για τις δύο παρουσιάσεις, αλλά αυτό προβλέπει η διαδικασία. Αυτοί είναι οι κανόνες που ισχύουν. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ο κύριος Σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευγενική πρόσκληση. Είναι τιμή μου να σας μιλήσω εδώ απόψε και να σας παρουσιάσω τα πορίσματα της μελέτης που διεξαγάγαμε για αυτήν την ε, Επιτροπή για το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, στην Ήπεθρο. Ο κ. Μπεντσού από την Αυστριακή από τον Αυστριακό Οργανισμό για την Ανάπτυξη της Υπέθρου και εγώ ίδιος από την CCR θα κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε είναι πρώτα απ' όλα τι είχαμε να φέρουμε εις πέρας, μετά κάποια από τα πορίσματά μας, κάπως συνοπτικά, και μετά συμπεράσματα όσο το δυνατόν πιο ε, σαφή. Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να κάνουμε μία ανάλυση της συνεισφοράς της ε, ΚΑΠ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ήπεθρο στην Ευρώπη. για να τροφοδοτήσουμε και την ε, έκθεση της νομοδότης ιδίας πρωτοβουλίας για την οποία θα μιλήσετε στη συνέχεια. Εδώ είδαμε το, Είδαμε το δυναμικό της ΚΑΠ να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο. Δηλαδή τα καθαρά δεδομένα που μπορεί να διαθέτουμε αριθμητικά, αλλά και τα συμπεράσματα που μπορέσαμε να διεξαγάγουμε. Επίσης κοιτάξαμε σε ποια κράτη-μέλη και σε ποιες περιοχές του η ΚΑΠ υπήρξε πιο αποτελεσματική στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και στραφήκαμε μετά στο ε, ζήτημα του κατά πόσο η ΚΑΠ επηρεάζει την απασχόληση στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα αντιστοίχως. Αυτό που χρειάστηκε να κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο, μια τριγωνική μορφή με τα πορίσματα στο τέλος, τα στοιχεία στην πάνω γωνία και προσπαθώντας να δούμε τα ζητήματα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η πρώτη είναι να δούμε τα στοιχεία της βιβλιογραφίας, στα οποία δεν θα μπω καταλέμε με λεπτομέρειες, μετά να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση των ε, καθαρών δεδομένων και των στατιστικών πληροφοριών που διατίθενται για το θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε δεν θέλαμε να εξεύρουμε κάποιο νέο μοντέλο, ένα παράδειγμα και μετά κοιτάξαμε αναπερίπτωση κάποιες ε, ε, υποθέσεις των κρατών μελών σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε επίπεδο περιφερειών ή επαρχιών για να δούμε τι επιπτώσεις υπήρξαν και εν τέλει όλα αυτά τα στοιχεία να τα εκφράσουμε σε συμπεράσματα. Όπως υπόθηκε ο στόχος μας ήταν να εξετάσουμε τη βιβλιογραφία κατά λεπτός. Και αυτό το κάναμε συστηματικά με επιστημονική προσέγγιση. Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τα στοιχεία από το 92 και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ετερογενή. Δηλαδή, ο αντίκτυπος της ΚΑΠ ω προ την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση ήταν θετικό ή αρνητικό, ανάλογα με διαφορετικού παράγοντε. Πρώτα απ' όλα, τι διαφορέ μεταξύ των γεωργικών κλάδων των κρατών μελών, έπειτα τα διαφορετικά εργαλεία πολιτικής που χρησιμοποιήθηκαν κατά, καιρού, κατά καιρούς και μετά η διαφορετική μεθοδολογία που χρησιμοποιηθηκαν κατα καιρου και μετα η διαφορετικη μεθοδολογια που χρησιμοποιηθηκε για να καταλήξουμε σε διάφορες εκτιμήσεις εφόσον δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο συμπέρασμα από όλη αυτή την έξαταση της βιβλιογραφίας, μπορούμε να δούμε πώς πολλοί συντάκτες μελετών συμφωνούν ότι ο βασικός αντίκτυπος της ΚΑΠ ήταν να διατηρήσει παρά να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι η ΚΑΠ εξυπηρέτησε στο να μειωθεί το ποσοστό εξόδου εγκατάλειψης του γεωργικού κλάδου από τους γεωργούς. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου κάποιες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν, η βιώσιμότητά τους μακροπρόθεσμα δεν ήταν και πολύ βέβαιη. Δηλαδή πολλές, παρόλα αυτά, εξατμίζονταν μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο μελέτης. Αυτό είναι ακόμη πιο σαφές, αν δούμε τις δημοσιεύσεις, που προσπάθησαν να προβλέψουν εκ των προτέρων το μέλλον της ΚΑΠ ε, όλος ιδιαιτέρως τις διαδικασίες απελευθέρωσης που θεωρήθηκε ότι θα μειώσουν τις δυνατότητες εργασίας των οικογενειών ή των εξωτερικών συνεργατών. Οι αρνητικές τώρα συνέπειες μπορεί να είναι άμεσες ή και έμεσες. Οι δρόμοι δράσεις της ΚΑΠ είναι το εισόδημα, το κεφάλαιο και οι επενδύσεις. Αυτά έχουν διαφορετικές ε, επιδράσεις ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης, της οικογενειακές λόγου χάρη. Η βασική οδός με την οποία λειτουργεί η ΚΑΠ είναι το εισόδημα. Όταν οι οικογένειες έχουν ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα, λιγοστεύουν οι πιθανότητες, λιγοστεύουν τα κίνητρα να εγκαταλείψουν αυτόν τον κλάδο. Από την άλλη όμως, οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής, γεωργικής παραγωγής λαμβάνουν τέτοια στήριξη που εντατικοποιούν την παραγωγή τους, συμπυκνώνουν την ε, παραγωγή και τις μεθόδους και τελικά είναι θετικός ο αντίκτυπος για την παραγωγικότητά τους και το εργατικό τους δυναμικό και το πώς τα αξιοποιούν. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζονται και λιγότερους εργάτες. Τώρα ως προς την ανάπτυξη της υπαίθρου, η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι τα προγράμματα ανάπτυξη της υπαίθρου που ήταν πιο αποτελεσματικά ήταν αυτά που είχαν να κάνουν με συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή τον αριθμό των θέσεων απασχόληση που δημιουργήθηκαν. Όμω, λάβαμε υπόψη τα προγράμματα ανάπτυξη τη υπαίθρου, γιατί συνήθω είναι σχεδιασμένα να δημιουργήσουν νέε ευκαιρίε απασχόληση στι γεωργικέ οικονομίε συνολικά. Οπότε οι γεωργοί μπορούν να αποφασίσουν εάν θέλουν να αλλάξουν τομέα δραστηριότητα. Όπως τον τομέα της ε, φιλοξενίας, ας πούμε, ή τον ε, τουριστικό. Τέλος, η βιβλιογραφία ε, ασχολείται με πολλά διαφορετικά στάδια μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Μεταξύ αυτών, οι περισσότερες μελέτες συγκεντρώνονται στη μεταρρύθμιση του 2003. Αυτό σημαίνει ότι μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της μεταρρύθμισης, όπως την μελετήσαμε, ήταν η αποσύνδεση. Η μεταρρύθμιση αυτή μαζί με την αποσύνδεση θεωρήθηκε από πολλούς μελετητές ότι ήταν αρνητική. Δηλαδή, όταν οι γεωργοί ελάμβαναν στήριξη ασχέτως του όγκου παραγωγής τους, είχαν και λιγότερα κίνητρα για να εργαστούν παραπάνω στα χωράφια. Αυτή, ε, αυτό το, αυτός ο επιπλέον χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους κάποιες φορές χρησιμοποιείται για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με άλλες μη γεωργικές δραστηριότητες. Ο Μπέντορα. Ευχαριστώ. Να δούμε τη στατιστική ανάλυση όπου δοκιμάσαμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ε, για να συνδυάσουμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση με διαφορετικούς τρόπους. Προσπαθήσαμε από τη μια να δούμε την συνεισφορά της ΚΑΠ, όπως είδατε και στη διαφάνεια, ε, δεν σας εκπλήσει, το γνωρίζετε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Καταρχήν, οι δαπάνες τη ΚΑΠ αυξήθηκαν ε, στο διάστημα 2000-2014 με μία τάση σταθεροποίησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και υπήρξε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης της υπαίθρου. Το βλέπετε στις ε, ανοιχτές πράσινες στήλες. Αυτό λόγω των άμεσων ε, βοηθειών πληρωμών που όλοι γνωρίζουμε. Είναι προφανές αυτό το συμπέρασμα. Όμως προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και τις διασυνδέσεις ή για να το πω αλλιώς τους αλληλοσυσχετισμούς μεταξύ των γεγονότων αυτών και του, της παραγωγής της Γεωργίας, των αποτελεσμάτων της Γεωργίας. Βλέπετε εδώ τι δόθηκε αν ε, εκτάριο ε, στη γη ε, την καλλιεργούμενη. Το βλέπετε με πράσινο στα αριστερά. Βλέπετε οι παραδοσιακά γεωργικές χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία να βρίσκονται και πάλι σε ηγετική θέση. Ενώ η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σε άλλη θέση. Είναι βέβαιος κάπως προεκλανητικό αυτό το γράφημα, διότι δείχνει σωρευτικά τι χρηματοδότηση δόθηκε ένα εκτάρι μεταξύ του 2007 και 2013. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι πολλά νέα κράτη-μέλη δεν χρηματοδοτούνταν ακόμη, δεν συμπεριλαμβάνονταν στον υπολογισμό αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Εάν τα βλέπαμε σε μικρότερα, πιο τεμαχισμένα χρονικά διαστήματα όλα αυτά τα στοιχεία, θα βλέπαμε διαφορές μεγαλύτερες. Αλλά το εντυπωσιακό είναι τι χρηματοδότηση δόθηκε και τι ε, παραγωγή υπήρξε. Δηλαδή η ανάπτυξη στην ίδια περίοδο, 2007 με 2013, και με αιτήσιες εργατομονάδες, εργα... είναι αυτό που βλέπουμε με το, κόκκινο, το... με το σκούρο κόκκινο μείωση των εργατικών μονάδων ανά εκτάριο και ανά λεπτό ευρώ. Στο πράσινο βλέπετε την ε, αύξηση. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη ο όγκος εργασίας που πήγε στην Γεωργία μειώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Ιδίω στην Ιταλία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και μόνο να αυξήθηκε σε πολύ μικρά μέρη της ε, Ευρώπης όπως η Ουγγαρία, η Κροατία, και κάποιες περιοχές της Σκοτίας και της Ιρλανδία και άλλη της αποτελεσματικοτητας τη αποδοτικότητα της γεωργιας αλλα εξυπακουει επισης μειωση στην χρηση του ίδιου νομίσματος. Ταυτόχρονα Ως πώς την απασχόληση αυτή καθεαυτή, δεν θα σας τα δείξω, αλλά τα λέει η έκφραση. Η ίδια εικόνα διαμορφώνεται, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη η απασχόληση στη Γεωργία μειώθηκε. Μειώθηκε για όλα σχεδόν τα κρατημέλη μεταξύ του 2008 και 2014. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Κροατία. Η Λετωνία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Η Ρουμανία μάλιστα είναι ειδική περίπτωση, διότι είχαμε αύξηση 20% στην απασχόληση. Δηλαδή τελείως κόντρα στο ρεύμα. Η άλλη εικόνα που θέλω να σας δείξω είναι η σχέση μεταξύ της χρηματοδότησης, δηλαδή του τι δώσαμε στην ΚΑΠ, ως πληρωμές της ΚΑΠ, και το τι αποτέλεσμα πήραμε. Το βλέπετε από τη μια με πράσινο, οι συνεισφορές ε, σωρευτικά στους διάφορους πυλώνες της ΚΑΠ με πράσινο, με κόκκινο σκούρο μάλλον, βλέπουμε τις άμεσες πληρωμές, με ανοιχτό κόκκινο βλέπουμε τις πληρωμές ανάπτυξης της υπαίθρου, Βλέπουμε ότι περισσότεροι δικαιούχοι, αυτοί που πήραν τα περισσότερα ήταν Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα. Αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα τους πρόλαβε και η Πολωνία. Αυτό είναι το συνολικό ποσό. Διότι αυτές είναι μεγαλύτερες, πιο βαριές γεωργικές χώρες της Ευρώπης. Στα δεξιά κάτω στη γωνία βλέπετε το αποτέλεσμα σε σχέση με τις συνεισφορές που δόθηκαν ως προς τις πληρωμές. Αυτό που μας εκπλήσει είναι ότι στην πορτοκαλιά στήλη που βλέπουμε στατιστικά τον όγκο παραγωγής, τα αποτελέσματα της γεωργίας, αύξηση παντού στην Ευρώπη ασχέτως του τι πήρανε. Εάν πήραν περισσότερη ή λιγότερη χρηματοδότηση οι διάφορε χώρε. Ενώ οι πράσινε στήλε τι σα δείχνουν. Σα δείχνουν το αποτέλεσμα ω προ την χρησιμοποιούμενη ευρωκροτική γη, τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων και τη συνεισφορά εργατικού δυναμικού στη Γεωργία. Βλέπουμε παντού αυτοί οι αριθμοί να μειώνονται. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχουμε μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων και αύξηση του μέσου όρου μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, καθώς και μείωση συνολικά της απασχόλησης στη Γεωργία εν τέλει. Αυτά ήταν απλώς πορίσματα, κάποια πορίσματα, κάποια μικρά συμπεράσματα από την στατιστική μας ανάλυση. Όμως αυτά τα συνοδεύσαμε με την αναπερίπτωση μελέτη κάποιων υποθέσεων σε κάτι μέλη. Δεν θα μπω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά είναι σημαντικό να επισημάνω αυτό που είπε και ο Μάουρο, ότι η εξέταση της βιβλιογραφίας τι έδειξε, ότι ό,τι διαπιστώσαμε από εκεί αποδείχθηκε και από τις ε, αναπερίπτωση μελέτες. Δηλαδή, Τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι η ενίσχυση δόθηκε όχι για να δημιουργήσουν νέε απασχόλησης αλλά για να συντηρήσουν αυτές που ήδη υπήρχαν. Και κάποιες φορές, μάλιστα ήταν και αρνητικός παράγων η χρηματοδότηση, δηλαδή η απασχόληση, θεωρήθηκε ότι απειλήθηκε από τον πρώτο πυλώνα λόγω της μεγάλης αποσύνδεση, της μεγάλων τάσεων αποσύνδεση και της μεγάλης στροφής προς την αγορά. Δηλαδή εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα της γεωργίας. Και ταυτόχρονα μείωση της απασχόλησης. Από την άλλη, όπως υπόθηκε και στην εξέταση της βιβλιογραφίας, τα προγράμματα της ανάπτυξης της υπαίθρου θεωρήθηκαν ως πραγματικά δημιουργώντα θέσεις απασχόληση, αλλά όχι απλώς στο γεωργικό κλάδο και σε άλλους τομείς της υπαίθρου, δηλαδή στις αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στα κάτι μέλη. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι μέσα από, την αναπερί... από τις αναπερίπτωση μελέτες διαφαίνεται μια ισχυρότατη τάση στα κράτη-μέλη. όπου έχουμε μεθόδους επικερδής και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς γεωργικούς κλάδους, στην Ισπανία λόγω χάρη, στην, ε, στα, στα ή σε άλλες περιπτώσεις στην Ιρλανδία, στο γαλακτοπαραγωγικό τομέα, εκεί θεωρήθηκε περισσότερο εμπόδιο η ΚΑΠ, πρόσκομα, διότι δεν τους άφηνε να αξιοποιήσουν τις αγορεστικές τους δυνάμεις. Αλλά υπήρχε και η τάση, ιδίω για αυτές τις πολύ ανταγωνιστικές οικονομίες, όπως ε, την παραγωγή των γαλακτοκομικών, των φρούτων, των λαχανικών υπήρχε η τάση να καταλείπεται η γεωργία. Σε κράτη-μέλη όπου οι συνθήκες παραγωγής δεν είναι πολύ ευνοϊκές. Θα πάω κατευθείαν στα συμπεράσματά μου τώρα. Πρώτο συμπεράσμα που μπορούμε να αντλήσουμε από όλα αυτά τα απορίσματα είναι ότι ως προς το ερώτημα, ποιο είναι τελικά το αποτέλεσμα της ΚΑΠ και ποιον αντίκτυπο είχε στην απασχόληση στα διάφορα, στους διάφορους κλάδους της γεωργίας, πρώτον, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ως προς την αποσύνδεση είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση. Ενώ ο πυλώνας 2 μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος. Είναι ένα καλό παράδειγμα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Όπως όμως προείπα, όχι ακριβώς στον ακρεφνή γεωργικό κλάδο, αλλά σε άλλους κοντινούς τομείς, όπως την επεξεργασία τροφίμων, τον τουρισμό. Το δεύτερο συμπέρασμα παντλούμε είναι οι δυνατότητες της ΚΑΠ να μειώσει την απασχόληση στο γεωργικό κλάδο. Εδώ, όπως υπόθηκε από την εξέταση της βιβλιογραφίας και της περίπτωση μελέτες, ο πρώτος πυλώνας θεωρείται ως αυτός που διατηρεί θέσεις απασχόλησης αλλά δεν τις δημιουργεί. Και αυτό είναι ένα γεγονός που τελικά δεν έχει οδηγήσει σε ανατραφοδότηση του Γιώργου κλάδου με νέους γεωργούς. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τις διαφορετικές αλλαγές που ανέφερα, δηλαδή ο μέσος όρος μεγέθους εκμετάλλευσης αυξάνεται ή εργατικό δυναμικό ανά εκτάριο. Όμως ο, πυλώνας, ο δεύτερος πυλώνος δημιουργεί σίγουρα θέσεις εργασίας στο γεωργικό κλάδο, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει λοιπόν τάση διαφοροποίησης της γεωργίας, αυτό καταλαβαίνουμε. Το, το τελευταίο συμπερασμά μας για τη γεωγραφική διανομή και το ποια κράτη-μέλη ή περιοχές ήταν πιο αποτελεσματικοί στην δημιουργία θέσεων απασχόληση χάρη στην συμβολή τη ΚΑΠ, εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει σαφή απάντηση. Από τη μια, είναι κάπως δύσκολο να έχουμε ακριβή στοιχεία. Ό,τι εξήβραμε από τη μελέτη της βιβλιογραφίας ή από τις αναπερίπτωση μελέτες ήταν κάπως ετερογενές. Δεν ήταν σαφές σε επίπεδο περιφερειών τι έκανε η ΚΑΠ για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Οπότε, το μόνο που μπορούμε να πούμε με σαφήνεια είναι ότι δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για τον πρώτο πυλώνα και για τον δεύτερο πυλώνα είναι σαν την ε, σαν τη γάτα του Σέντιγκερ. Δηλαδή, πρέπει να δούμε πώς δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης λόγω των αναγκών της αγοράς. Δηλαδή, ξαφνικά ανοίγουμε ένα κουτί και τελικά βρίσκουμε το γάτα ζωντανή. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η τάση θα μειωθεί σε όλη την Ευρώπη λόγω των αναδιαφρώσεων και του περάσματος κονδυλίων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα που μπορεί κάπως να αντισταθμίσουν την απώλεια θέσεων εργασία. Και έτσι μπορεί να εξισορροπηθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου συνολικά. Μάλιστα και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μα τον κύριο Αντρέα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνωμονές μας για την παρουσία στην εκθέσεις τους. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πόσο δύσκολη υπόθεση είναι στην ιστορία της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για πρώτη φορά μας απασχολεί το θέμα της σχέσης της μεταρρύθμισης ΚΑΠ με την απασχόληση στην Ήπεθρο. Αναφερθήκατε στην απουσία αξιολόγησης κατά την σύνταξη της εκθέσης. Είχαμε και εμείς τις ίδιες δυσκολίες που επιδεινώνονται και επειδή η μελέτη προχώρησε παράλληλα με την κατάρτιση της έκθεσης. Μαζί με εσάς ανακαλύπτω και εγώ το περιεχόμενό της. Κατά κάποιο τρόπο πάντως ε, επιβεβαιώνει αυτά που θέλησα να καταγράψω και εγώ στην έκθεση για να οδηγηθούμε στη συζήτηση και την τελική βέβαια μορφή της έκθεσης που θα εγκριθεί τον Ιούλιο. Η απασχόληση και το ανέφερα δεν υπήρξε ποτέ κύριο μέλημα της κοινή γεωργικής πολιτικής από τις απαρχές της βέβαια. Τώρα και ενώ η διατροφική ασφάλεια τίθεται ε, σε διαφορετικούς όρους ως πρόκληση και ενώ η άνεργη είναι όλο και σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν μπορούμε συλλογικά να μην αντιμετωπίσουμε, να συζητήσουμε το θέμα του, της απόδοσης αυτού του 38% του προϋπολογισμού που αφιερώνει στην κυνηγεωρική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους απασχόλησης. Δεδομένου ότι και η απασχόληση είναι μία από τις 10 προτεραιότητες που έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα πρώτη σε σειρά ε, όπως την όρισε ο πρόεδρος Γιουνκέρ. Έτσι λοιπόν και με αυτές τις καταφάσεις, εάν θέλουμε την ΠΑΚ να την, κοιτά, την ΚΑΠ να την κοιτάξουμε όρους ε, θα πρέπει να την διατυπώσουμε σε τελείως νέες βάσεις. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι πρόκειται δηλαδή για μια πολιτική επιλογή στην οποία θα οδηγηθούμε εν τέλει. Η κοινή γεωργική πολιτική, όπως είπατε, έχει ένα μοντέλο επικρατή απαιτούν ε, εντατικής και παραγωγικά προσανατολισμένης γεωργίας, με μικρή δηλαδή παραγωγή θέσεων εργασίας, ε, προσανατολισμένο προς τις διεθνείς αγορές, χωρίς παραγωγή θέσεων και στη δεκαετία του 90 η προσέγγιση της γεωργίας προς τις αγοράς και οδήγησε σε μεγάλη φυτικότητα των τιμών και βλέπουμε πόσο δύσκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση σήμερα, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη αστάθεια ει βάρο και των εισοδημάτων, αλλά και των επενδύσεων και τη επασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όπω και εσεί διευκρινίζετε, προτείνεται αυτή η έκθεση σε δύο τμήματα. Στην μια ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιήσαμε εδώ στην Επιτροπή μα. Το πρώτο θα καλύπτει την ΚΑΠ στην τωρινή της μορφή με το κανονιστικό πλαίσιο και τα εργαλεία που μας προσφέρει. Και στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης θα ε, ορίζονται προοπτικές, θα περιγράφονται προοπτικές ε, σε σχέση με, τις, με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ για την απασχόληση μετά το 2020. Και αυτό ενώ το κείμενο δεν έπρεπε να περάσει τους 7.000 ε, χαρακτήρες σε έκταση, άρα έχω πολύ περιορισμένη έκταση κειμένου, αλλά είμαι βέβαιος και στηρίζομαι βέβαια στην υποστήριξη των συναδέλφων ότι με τι τροπολογίε θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το κείμενο αυτό και ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για του επόμενου μήνες και χρόνια. Στο πρώτο τμήμα τη έκθεσης, την τωρινή ΚΑΠ, που διατυπώνουμε κάποιες υποθέσει με βάση τα εργαλεία που έχουμε ζητήσει θέση αυτή τη στιγμή. Καταρχά, ενισχύεται η υποστήριξη, υπάρχει μάλλον η μελέτη της υποστήριξης της εγκατάστασης του νέου γεωργού που για πρώτη φορά εγγράφεται στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Ταυτόχρονα όμως θέλω, όπως είπατε και εσείς, να καλέσω όλα τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις για νέους γεωργούς που προβλέπει ο δεύτερος πυλώνας. Βλέπουμε τώρα ότι δεν αξιοποιούν όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη δυνατότητα, ώστε να εξασφαλίσουν την αναλλαγή στις γενναίες και την ανανέωση. Προτείνουμε λοιπόν να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο και τα μέσα για αναδιανομή των άμεσων επενδύσεων, τα άνωτα επίπεδα, και αυτό το λέω πάλι στην έκθεση, και να ε, επανεξετάσουν την αποσύνδεση. Γιατί η σύνδεση επέτρεψε να εγκαταλειφθούν κάποια είδη παραγωγής και να απεριμωθούν ορισμένες περιοχές πιο ευαίσθητες ε, ορεινές ε, ή πλαγιές βουνών. Μπορεί λοιπόν να συνεχιστεί με καλύτερες βέβαια προσπάθειες ε, προς την κατεύθυνση της αηφορίας. Το παρασύνισμα επίσης πιστεύω πρέπει να ξαναμελετηθεί εις βάθος με λιγότερη γραφειοκρατία για να έρθει πιο κοντά σε αυτή την γεωργική πρακτική που πολύ συχνά ο ίδιος ο Γεωργός παίρνει την πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσει. Επίσης, πρέπει να οργανωθούν οι κοινέ οργανώσεις αγορών με αποτελεσματικότερα μέσα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις, γιατί να στιγμής δεν εξασφαλίζεται αυτό, όπως το προτείνει η Επιτροπή. Προτείνουμε την έκθεση να προσανατολιστούμε περισσότερο προς μια γεωργία ποιοτική και με ανάπτυξη συστημάτων ποιοτικών τροφίμων σε άμεση συναφία με την περιοχή στην οποία αυτά παράγονται, αλλά και σε σχέση με τους παραγωγούς και εταίρους, είτε πρόκειται για ονομασίες προελεύσεως, γεωγραφικές ονομασίες ή βιολογικά προϊόντα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την περιοχή στην οποία παράγεται το προϊόν και πέραν αυτού έχουν να κάνουν και με την παραγωγή εκτός του τροφίμου και άλλων υπηρεσιών, πράσινης ε, χημίας, ε, διαφτήρηση βιοπικιλότητα, τουρισμό, προστασία περιβάλλοντος και προτείνω να αξιοποιηθούν τα σχέδια περιφερειακής ε, ανάπτυξης, μέσα από το δεύτερο πυλώνα δηλαδή, στοχευμένα για την αύξηση των θέσεων εργασίας, για την ανάπτυξη της απασχόλησης, γιατί βλέπουμε μερικές φορές τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης ότι εάν μπαίνουμε σε όρους απασχόλησης μπορούμε να παραγάγουμε προς τις εργασίας, εάν την αφήσουμε κατά μέρος δεν τα καταφέρουμε. Και επίσης πρέπει να κοιτάξουμε τους συνδέσμους μεταξύ γεωργίας και λοιπόν παραγόντων στην ε, περιοχή, στην Ήμπεθρο, όπου βέβαια μπορούμε να εξασφαλίσουμε με τη συνεργασία της βάσης, με την bottom-up δηλαδή προσέγγιση, περισσότερες συνεργατικές σχέσεις και άρα παραγωγή θέσεων εργασίας. Και πρέπει να κοιτάξουμε επίσης πώς μία προσέγγιση σε πολλαπλά επίπεδα ε, απορρόφησης πόρων από ταμεία μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα φυστάμενα ταμεία για να ενισχύσουμε και την ύπεθρο και την απασχόληση. Για την περίοδο μετά το 2020 και μιλάω πιο γρήγορα σιγά σιγά, πρέπει να διατηρηθεί υποστήριξη στην κοινή γεωργική πολιτική. Ξέρουμε ότι αυτή τις επόμενες εβδομάδες θα απασχοληθεί για τον προπολογισμό. Ε, και είναι πολύ τόσο απαραίτητο κατά με να διατηρηθεί η στήριξη στη γεωργία και γενικότερα την Ήπεθρο, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να ε, προχωρήσουμε στην επιλογή εκείνη, η οποία θα νομιμοποιήσει για τον πολίτη της κοινής πολιτικής, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο θα έλεγα μεταξύ γεωργίας και ευρωπαϊκής κοινωνίας με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασία πιστεύω ότι θα έχουμε κερδίσει αυτό το κρίσιμο στοίχημα. Εάν λοιπόν η απασχόληση στις περιοχές υπαίθρου μπορεί να προχωρήσει, εάν θέλουμε να καταστεί στόχους μας, πρέπει να ξαναδούμε το μοντέλο της γεωργικής ανάπτυξης, τις δομές βεβαίως των εκμεταλλεύσεων, αλλά και τους τρόπους της παραγωγής, τα είδη της παραγωγής. Λέμε ότι πρέπει να, να παράγουμε περισσότερα. Ναι, αλλά πάνω απ' όλα κατά καλύτερο τρόπο και κατά τρόπο αηφόρο. Αλλαγή λοιπόν στα μοντέλα παραγωγής, αλλαγή τρόπου σκέψης και νέες εξελίξεις που απαιτούνται ώστε να συνδυαστούν οι οικονομικές, οι οικολογικές και οι κοινωνικές ε, αλλαγές νοοτροπίες για να αντιμετωπίσουμε την απέτηση της ανταγωνιστικότητας βεβαίως θα πρέπει να πούμε και τι εννοούμε ως ανταγωνιστικότητα γιατί μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να δώσουμε απαντήσεις στην ανάγκη για αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο και το περιβαλλοντικό, το οικολογικό συμβόλαιο, στις απαιτήσει της ε, εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οι μικρές και μεγιστές επιχειρήσεις που γενικά παράγουν περισσότερη προσθεμένη αξία και ε, δημιουργικότητα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε για καλύτερα και πιο ποιοτικά συστήματα παραγωγής και τροφίμων αλλά και ε, υπηρεσιών και προϊόντων εκτός των τροφίμων. Πρέπει λοιπόν να στραφούμε σε νέες λύσεις, να έχουμε μέσα διαχείρισης των αγορών προσαρμοσμένα να επαναπροσδορίσουμε μηχανισμούς ε, ρύθμισης, διαχείρισης, διαμεσολάβησης, να αντιμετωπίσουμε την ποιητικότητα των τιμών που αποβαίνουν εις βάρος και των τιμών ε, στον καταναλωτή και της απασχόλησης. Πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή την πρόταση για την αποσύνδεση με μέτρα είτε πρόληψης των κυκλικών τάσεων είτε ε, ασφαλιστικού χαρακτήρα και η ανάπτυξη μέτρων όπως το ΣΥΛΕΛΔΙ ή το LEADER να, μπορούμε να πούμε ότι αφού απέδειξαν τα προγράμματα αυτά την, την αποδοτικότητά τους θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο και να πτυχθούν περαιτέρω. Πρέπει να δώσουμε έμφαση και κίνητρα για τις επενδύσεις που θα παράγουν τις εργασίες, να διαφυλάξουμε και αυτό είναι απαραίτητο τώρα για τη διασφάλιση της απασχόλησης τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται στην Ήπειθρο και για να κλείνω μετά το 2020 πρέπει να αποφύγουμε τις ε, ε, δογματικές αγκυλώσεις, να αναλογιστούμε μια πλήρη αναδιάρθρωση ακόμη και των τριών πυλώνων. Δεν πρέπει να διστάσουμε να προχωρήσουμε προς μια πραγματική κοινή πολιτική, με τους πυλώνες της ΕΣΤΟ, αλλά ταυτόχρονα και μια δημόσια πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου. Αυτή είναι η άποψη. Σας ευχαριστούμε κύριε Ανδρία. Ήταν εκτενής η παρουσίαση. Νομίζω ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν το λόγο το δήλωσαν. Εκπονήσαμε τον κατάλογο. Πρέπει να ξέρω πόσοι θα μιλήσουν για να κατανείμω και το χρόνο το διαθέσιμο. Θα έλεγα δύο λεπτά στους και ηγητές, δύο λεπτά στους συντονιστές και οι υπόλοιποι από ένα λεπτό ο καθένας. Πρώτα που είναι ο από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες γενικές και κάποιες πιο ειδικές παρατηρήσεις και σχόλια για το σχέδιο έκθεσης. Θεωρώ καταρχήν ότι η κοινή γεωρική πολιτική ε, με το δεύτερο πυλώνα δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα ανεργίας στην Ήπεθρο και ενεργεία κυρίως μαστίζει ε, την Υπεθρό, αλλά αυτό είναι μόνο ένα τμήμα. Τι σημαίνει αυτό το νεύμα κύριε Πρόεδρε? Στην ε, Πολωνία 50% του πληθυσμού βρίσκεται στην Ήπεθρο και είναι 20% η γεωργία στην Ήπεθρο. Χρειαζόμαστε και κονδύλια από την πολιτική συνοχή για να λύσουμε την ανεργία στην Ήπεθρο. Επίσης, ε, αξιολογούμε τώρα τι μεταρρυθμίσει στην κοινή πολιτική. Και μάλιστα οι περιβαλλοντικές ε, αλλαγές υποφελήθηκαν, ε, τα περιβαλλοντικά θέματα υποφελήθηκαν από τις μεταρρυθμίσεις, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε και κοινωνικές συνέπειες θετικές από, τα, από τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πολύ δύσκολη επίσης είναι η κατάσταση στις γεωργικές αγορές. Πάλι διακοπή. problem Two minutes for the shadows and one minute for the others. For shadows we have no Ο χρόνος περνάει κύριε Καρινόφσκι, Το χρονόμετρο τρέχει. Να ξεκινήσω ή όχι ακόμη. Πρέπει να τα επαναλάβω όλα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας ακούμε κύριε Καλινόφσκι. Τότε να συνεχίσω αυτό που έλεγα, το τρίτο θέμα. Στο σχέδιο έκθεσης μιλούμε για την πολύ δύσκολη κατάσταση στις γεωργικές αγορέ, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία εν των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται και για το TTIP και με τη Μερκοσούρ. Αλλά ε, και με θέματα που αφορούν την Ουκρανία, την Αυστραλία. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικές, ε, υπερβολικά φιλόδοξες οι προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών αμμονίας και σίγουρα θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και σίγουρα θα επηρεάσουν και τις θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη τα θέματα που αφορούν την επιστημιστική αλυσίδα και να ενισχύσουμε σε αυτή την επιστημιστική αλυσίδα τη θέση των γεωργών, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που το αναφέρουμε συχνά. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε διεξοδικά για το σημείο 20 του σχεδίου έκθεσης που αφορά τις οικονομ... τους κοινωνικούς όρους των εργαζομένων στην Ήπεθρο και το κοινωνικό dumping. Επίσης, ε, να δούμε αυτή την τάση που υπάρχει επανεθνικοποίηση της γεωρικής πολιτικής. Ε, έχουμε αφενός το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που ενισχύεται από τις, ενισχύ, από τις της συνθήκης για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς γεωργικού εισοδήματο στους Ευρωπαίους γεωργούς αφενός και αφετέρου όλο και παρεκκλίνουμε από τις ρυθμίσεις της αγορές και όλο και περισσότερο α, ανοιγόμαστε προς τις εισαγωγές και εισάγουμε προϊόντα από τον κόσμο ολόκληρο. Θα πρέπει να πούμε ευθαρσώς ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είτε θα περιοριστούμε στις ευρωπαϊκές με ε, ρυθμίσεις, είτε θα πούμε ναι στην ανοιχτή αγορά. Αλλά και το ένα και το άλλο ταυτόχρονα δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μίλλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως τους δύο εισηγητές και τους συντάκτες της μελέτης. Βεβαίως, πολλά ακόμα πρέπει να διευκρινιστούν εν γέννη. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα, δεν είχαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα πλήρη εικόνα των 28 κρατών μελών και τα απαραίτητα λεπτομερή δεδομένα. Πράγμα το οποίο θα ήταν για μένα το, το ε, απαραίτητο, δηλαδή να έχουμε μια πολύ καλή βάση δεδομένων για να μπορέσουμε να συζητήσουμε την υπόθεση αυτή ε, εντατικά. Με την υποστήριξη λοιπόν, το ε, η υποστήριξη της απασχόλησης είναι απολύτως απαραίτητη και κατεπηγόντως αναγκαία. Στην έκθεση δεν βλέπουμε επί της ουσίας ιδιαίτερη τέτοια τάση. Λέει βέβαια η έκθεση πως μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των θεσμών εργασία στην Ήπεθρο με την ΚΑΠ, αλλά δεν βλέπω να αναφέρονται συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα έχουμε μια ΚΑΠ με ένα ε, μοντέλο δύο πυλώνων, το 30% όπως λέει και η έκθεση των θέσεων εργασία προκύπτει από τον πρώτο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα επίσης προκύπτει ένα καλό δυναμικό, ένα, μια καλή ε, δυνατότητα δημιουργία της εργασίας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε με πιο σαφείς όρους και εντατικούς όρους το πώς ακριβώς θα κάνουμε ε, για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και μια και λαμβάνω το λόγο σχετικά Απροετοίμαστε για το άνοιγμα μιας γενικής συζήτησης σε σχέση με μια αναθεώρηση της ε, ΚΑΠ και ανατροπής ε, του συστήματος. Νομίζω ότι είναι ίσως υπερβολική αυτή η προσέγγιση. Ε, χρειάζεται βεβαίως βελτίωση μέσα στο δεύτερο πυλώνα. Έχουμε κάποιες δυνατότητες που προσφέρει η γεωλογική πολιτική όπως έχει αυτή τη στιγμή. Αυτές τις δυνατότητες πρέπει συγκεκριμένα να αξιοποιήσουμε και θα πρέπει νομίζω να πούμε ξεκάθαρα πως η κοινή γεωργική πολιτική έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες για τις πιο ε, μειονεκτικές περιοχές, αλλά και ε, το ίδιο πράγμα έχει εξασφαλίσει και η αποσύνδεση και αυτή είναι η δική μου εμπειρία από τη Γερμανία. Ευχαριστώ κύριο Σκάρθη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πολλοί προλαλήσαντες ε, στάθηκαν στα κεντρικά σημεία της έκθεσης. Και θα ήθελα ευκαιρία να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονές μας και τον ε, εισηγητή μας για τη συνεισφορά τους. Μπορεί η Γεωργία από μόνη της να μην είναι ο σημαντικότερος εργοδότης σε όλες τις περιοχές, αλλά κυρίως στις περιφερειακές περιοχές, περιφέρειες, είναι η, ο κινητήριος μοχλός της τοπικής οικονομίας. Και ε, πολλές περιφέρειες ε, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τη Γεωργία. Θα πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να διαφυλάξουμε ε, μετάβλητο τουλάχιστον τον γεωργικό προπολογισμό και να διαφυλάξουμε και τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς. Επίσης, αν συμφωνήσουμε σε αυτά τα δύο σημεία που προανέφερα, θα πρέπει να δούμε πώ θα αναδιανύμουμε τα κονδύλια για να υλοποιήσουμε αυτού του στόχου. Γιατί είναι σαφέ κατά τη γνώμη μου ότι για να ευνοήσουμε τις τοπικέ οικονομίες ιδιαίτερα στις α, ε, α, ε, περιφερειακές ζώνες, που μεγάλο τμήμα της απασχόλησης α, ε, εξαρτάται από τη γεωργία, εκεί είναι που οι πληρωμές της ΚΑΠ θα έχουν το, το μεγαλύτερο αντίκτυπο και οι, οι γεωργοί δυστυχώς από αυτές ακριβώς τις περιοχές που χρειάζονται λαμβάνουν τη χαμηλότερη αναλογία των ενισχύσεων. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να υπερασπίσουμε το γεωργικό προπολογισμό και τον προπολογισμό κυρίω του πυλώνα 1 τη γεωργική πολιτική και επίσης να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε συστηματική ανακατανομή ε, των πληρωμών, ώστε οι πληρωμές να πηγαίνουν όχι μόνο στους ε, χρήζοντες γεωργούς, αλλά και στις περιφέρειες ε, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτές τις πληρωμές από την ΚΑΠ. Και συμφωνώ με, το, με κάποιον προλαλήσαντα που είπε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις εμπορικές συμφωνίες και τον δυνητικό αντίκτυπό τους στις ε, ε, περιφερειακές αυτές ζώνες και στις αγροτικές όπως ε, ΤΙΤΙΠ, ΣΥΤΑ, Μερκοσούρ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί μπορεί να καταρρεύσει η γεωργία και να εξολαθευτούν πλήρω οι γεωργικέ εκμεταλλεύσει εξαιτία των αρνητικών συνεπειών των εμπορικών συμφωνιών. Ο κύριο Ροπέ. Δύο λεπτά και παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, θα πρέπει να δώσουμε απάντηση σε πολύ σημαντικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ε, τι εικόνα θα έχει αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό από το πρίσμα της ε, απασχόλησης, των νέων θέσεων εργασίας, αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε και όλα θέσεις απασχόλησης, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε βιώσιμες αυτές οι θέσεις εργασίας. Όχι μόνο να δημιουργήσουμε νέες, αλλά και να διαφυλάξουμε τις υφιστάμενες. Νομίζω ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα για όσους διαβιούν και εργάζονται στην Ήπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους γεωργούς μας για να παραμείνουν στην Ήπεθρο. Να βοηθήσουμε τον κόσμο που επαναλαμβάνω ζει και απασχολείται στην Ήπεθρο, όχι μόνο τους μεγάλους γεωκτήμονες. Επίσης, για το σύστημα πληρωμών. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ε, ως προς τις ενισχύσεις που λαμβάνουν οι γεωργοί τους. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία και μια ε, ισότητα. Επίσης, δεν υποστηρίζουμε δεόντως τους νέους ε, γεωργούς, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν οι νέοι την Ήπεθρο. Η Ήπεθρος αντιμετωπίζει πολλά κοινωνικά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την κατάσταση και στις χώρες προέλευσης και στις χώρες προορισμού και από κοινού να επιλύσουμε τα προβλήματα. Ένα άλλο σημαντικό σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Κατά τη γνώμη μου, οι ΟΤΑ θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο εμφανή ρόλο για στο δεύτερο πυλώνα ειδικά της κοινή γεωργική πολιτικής. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία για καλύτερη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των κονδύλιων. Ευχαριστώ κύριο Σουλάζο. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τις ε, συνέπειες ε, ε, των ρυθμίσεων αυτών στη γεωργία. Και πραγματικά έχω συγκλονιστεί και έχω αειδιάσει από έναν εμπειρογνώμονα που είπε ο κύριο Βιγκάνη, δεν κάνω λάθο, ότι χάρη στην ΚΑΠ θα διασφαλιστεί η απασχόληση Ήπεθρο. Είστε ψεύτη. Ε, ψεύδεστε κατάφορα. Δεν είναι η ΚΑΠ που βοήθησε να παραμείνουν θέσει απασχόληση ε, ε, στην Ήπεθρο. Στη δεκαετία του 50 είχαμε 10 εκατομμύρια θέσει εργασία, 31% του, ενεργού, του συνολικού ενεργού πληθυσμού. Και μόνο 4% έχουν απομείνει σήμερα ενεργό πληθυσμό στην Ήπεθρο. Και κανένα οικονομικό κλάδο δεν υπέστη τόσο δραματικά δραματική μείωση των θέσεων απασχόληση. Μπράβο, πείτε αν τολμάτε αυτά που μα δηλώσετε στους Γάλλου. Ήταν πολύ... Ήταν πραγματικά ψέματα, κατάφορα. Τα σε έπαιρνα με τις ντομάτες, αν τα λέγατε. Είχαμε το τελευταίε δεκαετίε πολύ μεγάλη μείωση των θέσεων απασχόληση, ενώ ο αριθμός των μεγάλων εκμεταλλεύσεων έχει μεγαλώσει, κάτι που είχε αρνητικέ επιπτώσει στην οικονομία, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και μεγαλύτερη απερίμωση και κατάληψη τη υπαίθρου. Νομίζω ότι η μόνη λύση για την επιβίωση των γεωργών είναι να ξεπεράσουμε αυτή την κοινή γεωργική πολιτική που κατέστρεψε τον ευρωπαϊκό και τον εθνικό γεωργικό ιστό. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε εξή ερωτήσει. Καταρχήν, κυριαρχία, εθνική κυριαρχία, υποστήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ε, επιστροφή της οικονομίας, ε, στήριξη των τοπικών οικονομιών, των μικρών δομών και φυσικά υποστήριξη της βιολογικής, οικολογικής γεωργίας και ίσως δημιουργία ε, αγορών μεταξύ των παραγωγών. Αυτό θα ήταν ένα σούπερ μάρκετ των παραγωγών μια πολύ καλή λύση. Οι εναλλακτικά προϊόντα, αυτά θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός νέου γεωργικού μοντέλου και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εξάρτηση που δημιουργείται τα, τις τελευταίες δεκαετίες. Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε όλα αυτά τα μέτρα ή θα αρκεστείτε και πάλι σε μια απλή και θεωρητική συζήτηση χωρίς όμως συγκεκριμένες και απτές προτάσεις. Κύριε Λοαζό, καλό ήταν α, να διαρωτηθείτε τι θα γινόταν στην Ήπεθρο αν δεν είχαμε την κοινή πολιτική ως προς τον αριθμό εργαζομένων και την απασχόληση. Ε, νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να τα πούμε αυτά και να μην τα λέτε στους εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Άγνιο, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω στη ζωή μου ολόκληρη παρατηρήσει τεράστια μείωση της ποιότητας της ε, απασχόλησης για τους γεωργούς από το δρεπάνι περάσαμε στη μηχανή του θερίσματος, από το τσουβάλι με το στάρι στις μεγάλες μηχανές, ε, της ε, ε, συσκευασίας από την εκρίζωση των ζυγανίων, ζυζανίων στη μαζική παραγωγή και χρήση ζυζανιοκτώνων. Εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον στη χώρα μου, αλλά και στις υπόλοιπες δεν νομίζω να υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί η απασχόληση. Εκτός και αν μιλήσουμε για τη βιολογική βέβαια παραγωγή και αυτό πάλι με βάση τις ανάγκες του καταναλωτή και εκεί πρέπει να δούμε τι είπαμε και χθε σε σχέση με το καλακτοκομικό τομέα. Ε, κοίταξα λοιπόν κάποιους τομείς που μπορούν να βοηθήσουν με την αύξηση της προσθέμενης αξίας ε, στο ε, προϊόν, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τη δασοκομεία. Αν πρόκειται λοιπόν να ρίξουμε δημόσιο χρήμα σε αυτούς τους τομείς, θα ήταν προτιμότερο ίσως να απαιτήσουμε να τηρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας αυτών που δεν υπάρχει και, να, και στη βελτίωση των προσβάσεων των οδικών σε αυτές τις περιοχές της Υπέθρου, γιατί έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τους ε, πολίτες που ζουν στις περιοχές αυτές, την διαμονή τους και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους, χωρίς να κάνουμε κάτι το ανόητο και το τεχνητό. Αν θέλουν να εργαστώ με τέτοιο τρόπο, βέβαια. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Εκπροσωπώ την κυρία Γκέρλινγκ και όδη της ομάδας μου που είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τους ομιλητέ για τις δύο αυτέ παρουσιάσεις. Υποστηρίζω την αναφορά σε ένα σύνδεσμο μεταξύ της Γεωργική και της ε, πολιτικής για την Ήπεθρο με βάση και το σχέδιο Γιούνκερ για μια ανάκτηση και ανάκαμψη της οικονομίας, ε, της γεωργικής αλλά και γενικότερα προς το στόχο της κατεύθυνσης δημιουργίας της εργασία. Χρειάζεται μια πιο εστιασμένη έκθεση που θα δίνει ένα σαφές απερίφραστο μήνυμα υπέρ της δημιουργίας της εργασίας στην Ήπεθρο και όχι μόνο στο γεωργικό τομέα ή την παραγωγή τροφίμων, αλλά γενικότερα. Κάτι το οποίο δεν πράττει η ε, έκθεση καθώς δεν έχει στοχευστεί ιδιαίτερα το στόχο ε, το στον πυλώνα 1. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε πιο ξεκάθαρα για την κάλυψη της περιφερειακής ανάπτυξης, για τις μεγάλες αποκλήσεις που υπάρχουν στην οικονομία στις, περιφ... στις περιοχές της Υπέθρου, στην υποστήριξη των ε, οικονομίων στην Υπέθρο που έχουν το δυναμικό δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξης. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους για τη χρήσιμη μελέτη. Θα συμβάλλουμε με τις τροπολογίες μας στη βελτίωση της εκθέσεως και πιστεύω ότι μπορούμε με τη συνεργασία αυτή να έχουμε καλές θέσεις εργασίας, περισσότερες θέσεις εργασίας. Ε, η υλοποίηση μιας πολιτικής για την Ήπεθρο μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μεταβλητές, να μας δώσει απαντήσεις για την ε, δημιουργία λάθος εργασίας και σε σχέση με τον πυλώνα 2 και νομίζω ότι ήρθε, η ώρα να γίνει η, αν, ε, η επαναμελέτη των ε, ενισχύσεων που προβλέπονται γιατί οι ενισχύσεις από το σε νομικό ε, πλαίσιο για, το, για την ανάπτυξη πέθρου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Λαβετε το λόγο και στο όνομα της, ε, του σκιώδης συγητού ταυτόχρονα, ο κύριος Ντόρφμαν. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς τους ειδικούς μας. Εάν χαθούν θέσεις εργασίας από τη Γεωργία, αυτό νομίζω μπορεί να αφήλεται είτε σε ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη γεωργία, είτε στην κακή υπόσταση αυτών των θέσεων. Ωστόσο, εσείς το είπατε κάπως πιο κομψά, δηλαδή μας είπατε ότι η ΚΑΠ αποβαίνει όφελος των γεωκτημόνων τόσο ε, περισσότερο και όχι των γεωργών. Και έτσι τα κίνητρα που, είναι μέσα, που δίνονται μέσα από την πρημοδότηση δεν αποβαίνουν σ' όφελος της γεωργίας ε, αλλά των ε, ε, γεωκτημόνων. Θέλετε κάπως να μας το εξηγήσετε και να μας πείτε πού βλέπετε την προσέγγιση εκείνη η οποία θα μας επέτρεπε και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, αλλά και να μην χάσουμε θέσεις εργασίας. Και άλλη μια ερώτηση σε σχέση με τον πρώτο πυλώνα. Οι πληρωμές υπολογίζονται ανά με διαφορές μεγάλες αναπεριφέρεια και ίσως θα πρέπει να κοιτάξετε εάν η ΚΑΠ, εκεί που είναι υψηλότερε οι πληρωμές ανά εκτάριο σε κάποια περιφέρεια, έχει δώσει αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά για τη ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό δεν μας το δείχνουν οι στατιστικές προς το παρόν. Κάθε φορά, όπως είπαμε, οι πληρωμές εξαρτώνται από, τον αριθμό των, από την έκταση, από τα εκτάρια. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν αν βλέπετε κάποια τάση υπέρ των θέσεων εργασία προς τα άνω ή προς τα κάτω. Απάντηση. Από όχι, ο κύριο Μπράνη, συγγνώμη. Από τη συζήτηση αυτή νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε, να αποφασίσουμε τι μα ενδιαφέρει περισσότερο. Η θέση εργασία στη Γεωργία ή η θέση εργασία στην Ήπεθρο. Γιατί αυτό είναι το κέριο ερώτημα και εγώ θα ήμουν υπέρ των θέσεων εργασία στην Ήπεθρο. θέσει ε, οι οποίε μπορούν να διατηρηθούν και να ενισχυθούν ε, ε, και με πιθανολογούμενη μείωση των θέσεων εργασία. Και θα έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη ε, έμφαση στην, ε, στον αγροδασοκομικό τομέα και τη δασοκομεία. Από την άφηξη της ελεύθερης αγοράς στη Γεωργία, οι πολιτικοί έχουν μικρότερο ρόλο να διαδραματίσουν. Επαναλαμβάνω, έχουν μικρότερο ρόλο να διαδραματίσουν οι πολιτικοί με την ελεύθερη αγορά στη Γεωργία. Ο Γεωργός, ο πελάτης, ο καταναλωτή και ο προμηθευτή έχουν τον κύριο λόγο πλέον, ό,τι και να λέμε. Πρέπει λοιπόν η ΚΑΠ σιγά σιγά να μειώσει τον όγκο της, να συνιστά μικρότερο ποσό του ευρωπαϊκού προπολογισμού και δεν νομίζω ότι ο πολίτης Ευρώπης θα δεχθεί κάτι διαφορετικό. Όχι λοιπόν επιστροφή στις επιδοτήσεις, όχι επιδοτή στην στήριξη των τιμών, όχι επιστροφή στις, στα συστήματα των ενισχύσεων. Μπορούμε να κοιτάξουμε βέβαια τις πληρωμές για να κλείσει το χάσμα μεταξύ των περιοχών της υπαίθρου και των αναγκών του ε, πελάτη, γιατί ο πελάτης είναι και ψηφοφόρος, πρέπει να ξέρει λοιπόν τι θέλει από τη γεωργική εκμετάλλευση, τι θέλει από την ύπεθρο, τι είδους φρούτα θέλει να τρώει τη τελευταία ανάλυση. Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας για τις συνεισφορές τους και τον κύριο Ανδρία για τη δουλειά του. Προφανώς η Γεωργία, αλλά αυτό είναι γνωστό, χάνει εργαζομένους σε όλες τις δικές οικονομίες. Έχουμε ε, ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά με αύξηση της ανεργίας. Και βεβαίως η αύξηση της ανεργίας είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται. Μέσω από τη δουλειά του κυρίου Αντρία, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα συλλογισμό βάσει του οποίου η ΚΑΠ να μπορούσε να βοηθήσει σε αυτόν τον νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο με αυτά τα νέα και περίπλοκα προβλήματα που έχουν ε, αναδειχθεί. Μιλήσαμε χθε για τη διακύμανση, στις τιμές, για τις κρίσεις, τις επισητιστικές Πώ θα μπορούσε λοιπόν η να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των νέων προβλημάτων των γεωργών με μια νέα διαχείριση των κινδύνων, μια καλύτερη διαχείριση των τάσεων των αγορών. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Ξέρουμε πώ έχει αλλάξει η Αμερικανική πολιτική ε, προ αυτή την κατεύθυνση και με τόλμη θα έλεγα γιατί έγινε μια καμπή από τι άμεσε πληρωμέ σε συστήματα ασφαλιστικά, σε συνεταιριστικέ ε, μορφέ συνεργασία. Εδώ λοιπόν Εφόσον μιλάμε για ενδιάμεση αναθεώρηση, θα θέλαμε να τη δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση, όχι αυτή που τώρα προτείνεται και είναι αντίθετη από την επιθυμητά. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω στη σημερινή συζήτηση και καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω, κοιτώντα γύρω μου, ότι στα σημαντικά θέματα πολλοί συνάδελφοι λάμπουν δια τη απουσία του και τώρα έρχονται να μα μιλήσουν για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ε, θα ήθελα τουλάχιστον να δώσω απαντήσει σε συναδέλφου οι οποίοι είναι πάντα παρόντε εδώ. Ε, Θέσει εργασία στην Ήπεθρο. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι είναι πάνω απ' όλα εθνικό και περιφερειακό ζήτημα ζήτημα αρμοδιότητας εθνικής και περιφερειακής. Εγώ ξεκίνησα ως εκπρόσωπο σε τοπικό ε, συμβούλιο. Είχαμε στη Βαβαρία επίπεδο ανεργίας 50% σε μια περιοχή του κάτω Παλατινά του πολύ κοντινή στην Τσεχία με δυσμενείς γεωλογικές κλιματικές συνθήκες και ύστερα από 40 χρόνια κοινή γεωλογικής πολιτικής για να απαντήσω στον κύριο εκεί πέρα πίσω μπορέσαμε αξιοποιώντας ευκαιρίες που μας προσέφερε η Ευρώπη και αυτό λέω προς όλα τα νέα κράτη-μέλη ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο και να προχωρήσουμε με τελευταίες στατιστικές ανεργίας στην Γερμανία που έδειχναν για τη δική μου την περιοχή το χαμηλότερο ποσοστό, το δεύτερο χαμηλότερο, 1,2% Ανεργία για ολόκληρη τη Γερμανία. Μπορέσαμε δηλαδή σε μια φτωχική, φτωχή περιοχή με πάρα πολύ υψηλή ανεργία, να μειώσουμε πολύ την ανεργία, δηλαδή να δημιουργήσουμε πάρα πολλέ θέσει εργασία χάρη στην κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ, κύριο Γιάρ. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω μια παράκληση Είπε ο κύριο Μίλλερ ότι αν βάλουμε πολλά θέματα μέσα στι προτάσει θα χρειαστεί πολύ καιρό όπω έγινε με την προηγούμενη κοινή γεωργική πολιτική, με την προηγούμενη μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική που χρειάστηκε χρόνια για να ε, επεκταθούμε σε όλα τα ζητήματα. Καταρχά, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προ την έκταση του ζητήματο και επίση θα ήθελα για του εμπειρογνώμονε. Όταν γίνεται λόγο για τη δημιουργία θέσεων εργασία, αφενό μεν μιλούμε για ασφαλή, θέσει εργασία για το εργατικό μα δυναμικό, δηλαδή να μην είναι οι χαμηλότερε ε, δυνατέ αμοιβέ ε, και σε ασταθεί θέσει εργασία, μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τι αριστικέ. Και δεύτερον, θα πρέπει να είναι χρήσιμο το προϊόν που παράγουν αυτές οι, θε, οι θέσεις εργασίας, αυτοί οι απασχολουμένοι, γιατί διαφορετικά αποβαίνει βάρος της ίδιας της κοινωνίας ε, η όποια προσπάθεια. Μιλήσαμε για ε, συστήματα ανώτατο, κατώτατων ορίων, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ανώτατα όρια. Διαφορετικά δεν έχει κανένα, κανένα νόημα το σύστημα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνικός. Σε ό,τι αφορά την αύξηση της ανεργία ή τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης ε, στη Γεωργία και στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να το δούμε αυτό από κοινού με την επισητιστική ασφάλεια. Και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει να εξασφαλίσουμε δηλαδή αυτή τον επιστηστικό ανεφοδιασμό μόνο όταν έχουμε σημαντική μείωση της ανεργίας στη γεωργία. Και η σταθερότητα των θέσεων απασχόλησης είναι ζωτική σημασία για τη γεωργία. Οπότε οι μηχανισμοί στήριξη θα πρέπει να συνδέονται με την παραγωγή ένα εκτάριο. Γιατί ε, σε κάποιες χώρες και κυρίως στη Ρουμανία, σε ορισμένες περιφέρειες, οι επενδυτές ε, είναι κύριοι ε, των αγροτεμαχίων, αλλά ενδιαφέρονται μόνο για τις ενισχύσεις και όχι για την παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε την παραγωγή με τις ενισχύσεις. Ο κύριος Χόισλινγκ. Έφυγε ο κύριος ε, Άλμπερτ, ελπίζω να με... Έφυγε ο Άλμπερτ, ελπίζω να με ακούσει βέβαια μετά και να ενημερωθεί μια και έφερε το παράδειγμα της Βαβαρίας. Δεν έχουν όλες οι περιοχές την ίδια δυνατότητα για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας. Και πρέπει να αξιολογήσουμε εν τέλει εάν τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε έχουν διατεθεί κατά σωστό τρόπο. Και αν τα λεφτά που πληρώνει ο φορολογούμενο πηγαίνουν στη δημιουργία θέσεων εργασία. Αυτό δεν έχει απελευθερωθεί επαρκώ τα τελευταία χρόνια από τη Γερμανία μπορώ να δώσω παραδείγμα τη σύγκριση με την ανατολική με τα ανατολικά κρατήδια. Κατά 70% οι μεγάλοι γεωκτήμονε στην Ανατολική Γερμανία έχουν εξάρτηση από τι άμεσε ενισχύσει, ενώ οι μικρότερε επιχειρήσει Γερμανίας έχουν μικρότερο ποσοστό στι άμεσες πληρωμέ, άμεσε ενισχύσει, αλλά ε, γιατί δεν υπάρχει κριτήριο σε σχέση με την προσθεμένη αξία που παράγουν, πράγμα το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί στα κριτήρια της ε, ΚΑΠ Γιατί η παραγωγή οικολογική είναι προσθεμένη αξία και πρέπει και αυτό να υπολογίζεται. Κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Δε μίλησε για μια κατάσταση που ίσχυε πριν από 50 χρόνια στην Βαβαρία. Ο κύριος Φλάναγκας. Η κοινή αγροτική πολιτική, κατά την άποψή μου, έχετε δυνατότητα να δημιουργήσει θέσει απασχόληση και ένα από του τρόπους για να δημιουργήσει κανεί θέση σε αυτόν τον τομέα είναι οι γεωργοί να, κρατάνε τα ευρώ, ε, να μην κρατάνε τα ευρώ στις τσέπες του, αλλά να τα ξοδεύουν στην τοπική κοινότητα. Εάν συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση όπου έχουμε μέγιστες πληρωμές 150.000 ε, ευρώ που δεν θα ξοδευτούν βεβαίω τοπικά, αλλά όπω συνέβη στην Ιρλανδία και έχουμε πολλά αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό, θα δαπανηθούν στο να αγοράσει κανείς διαμερίσματα στην Κροατία ή ανά την Ευρώπη, αλλά σε καμία περίπτωση όχι σε τοπικό επίπεδο. Εάν περιορίσουμε το μέγεθο τη πληρωμή σε κάτι πολύ χαμηλότερο τι 150.000, τότε τα χρήματα αυτά μπορεί και να ξοδευτούν σε τοπικό επίπεδο. Εάν είχατε ακούσει τις λογικές προτάσεις ακόμη και μία κοντινή μου περιοχή, το Λίτρεον, θα είχε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια παραπάνω ε, ετησίως, 400 ευρώ για κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί της περιοχής και θα είχαν ξοδευτεί τοπικά, αντί να τα δίνουν ε, σε ανθρώπους με μεγάλους διοκτήμονες, το Λάρι Γκούντμαν, ο οποίος δεν ξοδεύει τα χρήματα του σε τοπικό επίπεδο, αλλά αγοράζει τζετ για την πάρτη του. Αυτό είναι το πρόβλημα της Γεωργίας και... Προφανώ, όταν κάποιο στην Ιρλανδία αγοράζει τζετ κατά αυτόν τον τρόπο, κάποιο άλλο θα πεινάσει. Κυρία Σένερα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνική. Από τη στιγμή που μιλάμε για θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ άμεσης και έμεσης απασχόλησης, γιατί η ισχύουσα ΚΑΠ καταστρέφει τις άμεσες θέσεις απασχόλησης. Και εδώ και μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συγκεκριμένη Επιτροπή Γεωργίας μιλούμε για τις ε, διαδοχικές κρίσεις που έπληξαν ε, το γεωργικό κλάδο και λέμε πως ε, πολλοί γεωργοί κλείνουν, χρεοκοπούν και εγκαταλείπουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Όσο και να επενδύουμε χρήματα στο δεύτερο πυλώνα τη ΚΑΠ και θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλου είδου ε, θέσει απασχόληση στη Ήπεθρο, δεν θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε αυτέ τι θέσει εργασίας αν ε, δεν διαφυλάξουμε τι άμεσε θέσει απασχόληση στη Γεωργία. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που παρατηρούμε εδώ και χρόνια ολόκληρα και αν δεν την αντιμετωπίσουμε, πολύ φοβάμαι ότι συνεχίσουμε τι επενδύσει, αλλά σε πολύ βραχυπρόθεσμες ε, και περασμένε θέσει απασχόληση, όχι μόνιμες. Στη Γαλλικία εδώ και πολλά, πολύ καιρό χάνουμε θέσει απασχόληση γιατί οι γεωργοί κλείνουν τι ε, αγροτικέ του εκμεταλλεύσει, σταματούν τη δραστηριότητα γιατί δεν μπορούν να συντηρηθούν ε, επειδή άλλοι χρησιμοποίησαν χρήματα του δεύτερου πυλώνα για να κάνουν τι δικέ του επιχειρήσει. Ευχαριστώ κυρία Σρέιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακολουθώ τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον και να θυμίσω στους συναδέλφους ότι χθε περάσαμε μια ολική συνεδρίαση μιλώντας για τις κρίσεις των κλάδων της Γεωργίας. Μετά μιλήσαμε για τον προπολογισμό το πρωί. Και το γεγονό παραμένει ότι κάποιοι γεωργοί είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που λαμβάνουν τέτοιες γενναιόδρες προσφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να στηρίξουν βεβαίω το περιβάλλον, για την οδηγία πλαίσιο για τα νερά. Ε, αυτό είναι μέρος της συνολικής εικόνας. Όμως το θέμα είναι, θα φροντίσουμε τα ένομα συμφέροντα των μικρομεσαίων γεωργών ή απλώς θα υποχωρούμε και θα τα παραχωρούμε όλα στη, στο δέλεαρ των μεγάλων επιχειρήσεων και της δικής τους ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν Πρέπει να δούμε ε, τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε με τη Γεωργία. Μιλάμε για βιοπικιλότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμένουμε συνεπεί σε κάποιου στόχου. Αυτό επιζητούμε. Μελέτε που να μα πούν τι γίνεται σε συγκεκριμένε χώρε. Ωραία. Άκουσαμε τώρα τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Λόγκο, μια και ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των αγοριτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τρόπο με τον οποίο η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο είναι σημαντικό θέμα, γιατί είναι θέμα που ευθυγραμμίζεται και με τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ανήγγειλε ο πρόεδρο Γιουνκέρ. Και χαίρομαι ιδιαίτερω για τη συμμετοχή μου σε αυτή τη συζήτηση. Η έκθεση του κυρίου Αντριέ πολύ σωστά επισημαίνει τον ε, ζωτικό ρόλο της κοινή γεωργικής πολιτικής που είναι βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο. Και η Ευρωπαϊκή Γεωργία χαρακτηρίζεται από 11 περίπου εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, που απασχολούν 22 εκατομμύρια ανθρώπους. Σημαντικό τμήμα βρίσκεται στην Ήπεθρο και σε συνδυασμό με την επεξεργασία τροφίμων και το λιανεμπόριο. Η Γεωργία δημιουργεί ένα κλάδο που εξασφαλίζει περίπου 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ε, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον την παρουσίαση της μελέτης ε, που ε, βλέπει μια αρνητική συνέπεια ε, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μετά τη μεταρρυθμίση της ΚΑΠ. Και οι πληρωμές που γίνονται με βάση τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ τώρα δεν έχουν, δεν έχουν σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά έχουν ε, σημαντικά θετικά αποτελέσματα έμεσα στην απασχόληση και στον ίδιο το γεωργικό τομέα, αλλά και σε συναφείς τομείς. Στο γεωργικό τομέα, οι άμεσες πληρωμές ε, ε, σταθεροποιούν το γεωργικό εισόδημα και μάλιστα σε ένα πλαίσιο με χαμηλές τιμές προϊόντων. Και μαζί με, τα, με τους μηχανισμούς αγοράς, τα εργαλεία της αγοράς ε, που ρυθμίζουν τις τιμές, ε, οι άμεσες πληρωμές αποτρέπουν ε, την απώλεια παραγωγής και θέσεων απασχόλησης. Και μάλιστα οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 46% του οικογενειακού γεωργικού εκμεταλλεύσεων μεταξύ 2005 και 2013. Θα πρέπει λοιπόν να παραβλέπουμε το αποτέλεσμα που έχουν και σε άλλους τομείς γενικώ ε, στην Ήπεθρο και όχι μόνο στη Γεωργία. Όπως σας είπα, ο επιστηστικός κλάδος απασχολεί πολλούς ε, ε, εργαζόμενους, αλλά γενικώ ο αγοροεπιστηστικός κλάδος έχει και έμεση θέση απασχόλησης στις μηχανές, για παράδειγμα, ή αγροτουρισμός. Επίσης, εποφελείται από τη σωστή διαχείριση το, του αγροτικού τοπίου και από τη σωστή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οπότε η συνέχιση της γεωργίας θα μας βοηθήσει να συντηρήσουμε θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Κάτι που σημαίνει ότι οι πληρωμές του πρώτου πυλώνα μπορούν να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δημιουργίας θεμελίων ε, τα οποία θα εδράζονται οι πληρωμές του δεύτερου πυλώνα σε συνδυασμό και με την αναπτυξιακή πολιτική. Οι επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, στι επιχειρήσει και στην καινοτομία είναι βασικέ δραστηριότητε που προτείνει ε, η πολιτική ανάπτυξη πέθρου. Και μάλιστα αυτό γίνεται και χάρη στην τεχνογνωσία και στη βελτίωση της παροχής ε, στοιχειωδών υπηρεσιών στην Υπεθρό. Μάλιστα, πολιτικές ανάπτυξη πέθρου βελτιώνουν όχι μόνο το γερικό τομέα, αλλά και άλλους ε, συναφεί τομεί και βοηθούμε και άλλες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον και να θάλουν. Όπως ε, δείχνει η έρευνα και τα πορίσματά της, ο δεύτερο πυλώνα τη κοινή γεωργική πολιτική είναι αποτελεσματικό στη δημιουργία θέσεων απασχόληση ε, στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να βρεθεί ε, βέβαια ε, ο σωστό εστιασμό από τα κράτη-μέλη και κάποια στρατηγικά προγράμματα ε, θα πρέπει να έχουν τέτοιου στόχου ώστε να μπορούν να φέρουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. 160 δισεκατομμύρια είναι οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην Ήπεθρο σε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς να υπολογίζουμε τι λαμβάνω από άλλους ε, κοινοτικού μηχανισμούς. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί σίγουρα και καταβάλουμε προσπάθειες για να προωθήσουμε και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να διευρύνουμε το πεδίο δραστηριοτήτων. Και μαζί με το πρόγραμμα ε, το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και με τη βοήθεια άλλων ε, διαρθρωτικών ταμείων προσπαθούμε να ενισχύσουμε την πολιτική ανάπτυξη στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα αρνητικά αποτελέσματα και φυσικά χρειαζόμαστε γι' αυτό την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών. Και η βελτίωση της χρήσης των κονδυλίων και αξιοποίησή τους ε, ε, είναι τοπική επιλογή και εθνική επιλογή. Θα πρέπει λοιπόν να κανονίσουμε από κοινού τις προτεραιότητες μετά από μία ε, αντικειμενική αξιολόγηση των αναγκών των ενδιαφερομένων. Τέτοια στοχοθετημένο προγράμματα είναι τα πιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει να αποδείξουμε και θετικά αποτελέσματα των πολιτικών μας. Ένας προϋπολογισμός που θα επικεντρώνεται σε αποτελέσματα ε, είναι απαραίτητος για να γίνεται σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων και να έχουμε και ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ποσοτικοποιημένους στόχους. Και να δούμε αν οι στόχοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες για τους οποίους έχουν χαρακτή. Επίσης, ε, νέες δυνατότητες ε, για το γεωργικό τομέα και την Ήπεθρο ε, προέρχονται και από την κυκλική οικονομία και από την βιοοικονομία. Όλες αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να στηρίξουν επίσης ε, το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ε, και το, τους στόχους της βιωσιμότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και κυρίες που τηρήσατε το χρόνο σας και τώρα για πέντε λεπτά το λόγο θα πάρουν οι εμπειρογνώμονες μας. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, θα ήθελα να εξηγήσω ποιο ήταν το βασικό μου μήνυμα από τη βιβλιογραφία που μελετήσαμε. Δεν είναι το θέμα ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης, όπως κάποιος ανέφερε. Και υπήρξαν και επικρίσεις σχετικά, αλλά αντιστρόφως να είμαι σαφής. Ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη Γαλλία υπήρχε μια σταδιακή διαδικασία συγκέντρωσης. Και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι ότι η ΚΑΠ επιβράδυνε αυτή τη διαδικασία για να περιορίσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι κάτι που ο κύριος Πάολο Ντεκάστρο ανέφερε, με το οποίο συμφωνώ 100%. Είναι σημαντική πτυχή οι πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων και αγροκτημάτων και σε επίπεδο πολιτικής. Τόσο, η διαχείριση του κινδύνου όπως ε, ενσωματώθηκε στον πυλώνα 2 δεν ε, χρησιμοποιήθηκε σωστά. Μόνο εννέα μέλη δεν εφήρμοσαν το μέτρο 17 εννοώ. με ένα μέσο όρο 1,4% του συνολικού προπολογισμού. Πολύ χαμηλό ποσό. Τέλος, το τελευταίο μου σχόλιο αφορά τον κύριο Φλάναγκαν. Είναι πολύ σημαντικό πώς δαπανώνται τα κονδύλια της ΚΑΠ από τους γεωργούς. Υπ' αυτήν την έννοια αυτό που προέχει είναι να σκεφτούμε του έμεσους, τις έμεσες επιπτώσεις από τις δαπάνες. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν όπου οι γονεί δαπανούν το επιπλέον εισόδημά του στη γεωργία, συνήθω το δαπανούν για την εκπαίδευση, την παιδεία των παιδιών του. Αυτό οδηγεί συνήθω την νέα γενιά, την επόμενη γενιά, να ψάξει καλύτερε δουλειέ, άλλε δουλειέ εκτό γεωργικού κλάδου. Εάν δεν βρουν μια καλή δουλειά στο επίπεδο ε, που έχουν ε, επιτύχει, στο οποίο έχουν φτάσει σε μια περιοχή της υπαίθρου, Κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι ένα έμεσο αρνητικό αντίκτυπο του μεγαλύτερου εισοδήματο που έχουν οι γεωργοί. Ευχαριστούμε. Απλώς να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Μάουρο. Εάν σας δώσαμε την εντύπωση ότι απλώς αναλύουμε για να πούμε ότι προφυλάχθησαν οι θέσει εργασία. Όχι. Εγώ το συμπεράσμα που σα είπα στι τελευταίε μου παρατηρήσει ισχύει. Η απασχόληση στη γεωργία μειώνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Όμω, με την παρουσίασή μου, και θα επανέλθω στο πρώτο ερώτημα και την πρώτη παρατήρηση που έγινε εδώ, εγώ στην παρουσίασή μου είπα ότι το θέμα είναι το ποσοστό αποδοτικότητας κιόλας της γεωργίας. Με τις στατιστικές αναλύσεις έδειξα ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η αποδοτικότητα αυξήθηκε. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, εάν αυτή, αυτή η αύξηση αποδοτικότητας και το επιπλέον εισόδημα που έχουν οι ιδιοκτήτες γης, όχι αναγκαστικά οι ίδιοι γεωργοί, Εάν αυτό οδηγεί στο αποτέλεσμα να ψάχνουν αλλού δουλειά οι άνθρωποι, χάρη σε αυτό το επιπλέον εισόδημα, δεν μπορώ να απαντήσω από τα πορίσματα που έχουμε. Το πρόβλημά μας, και αυτό μας οδηγεί στο επόμενο ερώτημα που επακολουθεί, είναι όταν στην κλίμακα μιας επαρχίας, μιας περιοχής υπάρχουν περισσότερες επιτυχίες, ή συσχετισμός της χρηματοδότησης και των θετικών επιπτώσεων στην αγορά εργασία. Αυτό παρεμποδίζεται από το γεγονό ότι δεν έχουμε στοιχεία αναπεριοχή για την χρηματοδότηση της ΚΑΠ στον πρώτο πυλώνα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και για εμά του ε, ερευνητέ και καταλαβαίνω και το επιχείρημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω γιατί δεν δημοσιεύουν τα πορίσματα αναπεριοχή για τον πρώτο πυλώνα για λόγου ασφάλεια των δεδομένων, όμω ω προ του ερευνητέ και τι μελέτε μα αυτό είναι πρόσκομα. Είναι ένα πρόσκομα που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε τελικά να καταλάβουμε τι γίνεται με τι χρονικέ σειρέ, να κάνουμε σωστέ συγκρίσει ε, και αναλύσει και δεν καταλαβαίνουμε πώς οι επιπτώσεις σε περιφερειακή κλίμακα, ε, οι επιπτώσεις της χρηματοδότησης, πώς ακριβώς επηρέασαν την κάθε περιοχή. Αυτά από την πλευρά του ερευνητού. Έχουμε κάποιους περιορισμούς. Συμφωνώ επίσης απολύτω με κάποια τα σχόλια ότι Καλύτερο θα ήταν να έχουμε πλήρη κάλυψη όλων των κρατών μελών και να συγκρίνουμε μεταξύ τους. Θα συμφωνήσω απολύτως αλλά δεν προβλεπόταν στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Ίσως όμως να είναι μια καλή παρατήρηση και να την σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εκπονήσει μια τέτοια μελέτη ή τέλος πάντων να την αναθέσει. Ε, συμφωνώ απολύτως ότι σε κάποιες πτυχές, ιδίως ως προς τις παραλυκόμενες συνέπειες της ΚΑΠ, και τις δευτερογενείς επιπτώσεις, για να τις πω έτσι, τις συνέπειες στην απασχόληση, την περιβαλλοντική προστασία ή τις επιπτώσεις από την οδηγία Natura 2000 και άλλες. Δεν τα αναλύσαμε κατά λεπτός, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να δούμε τις δευτερογενείς συνέπειες, για περιπτώσεις θετικών παραδειγμάτων ως προς την απασχόληση, διότι Υπήρξαν δυνατότητε απασχόληση κάτι παρακάτω στην αλυσίδα προστιθέμενη αξία. Δεν υπάρχει επιβολή όμω. Τόνισα και θα ε, κλείσω με αυτό. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι προφανώ αυτό που είπε και ο εισηγητή ισχύει. Θέλω να το υπογραμμίσω κι εγώ. Είναι μάλλον η κατάλληλη στιγμή χωρί να περάσουμε σε μια εντελεχή συζήτηση για την ΚΑΠ, είναι σίγουρα μια καλή στιγμή να σκεφτούμε αν η γεωργία μακροπρόθεσμα η γεωργία αυτή καθεαυτή είναι κάτι το επίκαιρο. Ή μήπω θα πρέπει να συσχετιστεί με άλλα θέματα όπως προστασία του περιβάλλοντος, η οικολογία και ένα ανάγκη για τρόφιμα. Ο κύριος Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και πιο σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω για μια φορά του ειδικού μα για τι απαντήσει του, όλου του συναδέλφου για την υψηλή ποιότητα τη συζήτηση. Αν το, το ερώτημα του κατά πόσον η απασχόληση θα πρέπει να μπει ω μέλημα μέσα στην τωρινή πάκαλα και στη μελλοντική, νομίζω ότι με τις σα όλε ε, δόθηκαν οι απαντήσει, Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία, πρέπει να καταστεί και προτεραιότητα μάλιστα ως στόχος, γιατί πολύ παλιότερα το πολύ πολύ να το λέγαμε ως ε, οξύμορο, ως αστείο, αλλά ε, ποτέ δεν συζητούνταν σοβαρά. Τώρα το ότι γίνεται λόγος για προτεραιότητα στην δημιουργία της συνεργασίας δείχνει ότι έχουμε αλλάξει και νοοτροπία και λαμβάνει θεμελιώδη σημασία η έκθεση. Γι' αυτό σας καλώ όλους να προσφέρετε με τις τροπολογίες σας ε, ε, στην έκθεση ώστε να μπορούμε να επισέλθουμε και στις ε, λεπτομέρειες και να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΚΑΠ, όπως μπόρεσα σε αυτή τη σύντομη έκθεση να την περιγράψω, αλλά και για μια μελλοντική ε, ΚΑΠ μετά από μια μελλοντική μεταρρύθμιση, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις, τους προσανατολισμούς που θα λάβει μια μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ποιότητα της ε, ανταλλαγής επιχειρημάτων και ευχαριστώ βέβαια όλες τις ομάδες που με στήριξαν, ιδιαίτερα δε τη Γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας για το στάδιο αυτό των εργασιών που ήταν ε, πολύτιμη συνδρομή της στην ε, κατάρτιση ενός κειμένου το οποίο όπως είπα θα πρέπει να εμπλουτιστεί με τις τροπολογίες επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Μέχρι 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Είδαμε ε, την συνέπεια της, τη συνέπεια της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής στην ε, Ήπεθρο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το θέμα της εδαφικής συνοχής δεν μπορούμε να το περιορίσουμε μόνο στο δεύτερο πυλόν. Επίσης, σημαντικό και ήταν η ανάλυση της κατάστασης όταν ε, το δε, ο δεύτερος πυλώνας ήταν η πολιτική συνοχής ε, και η περιφερειακή προσέγγιση. Επίσης, το θέμα της ε, απασχόλησης στην Ήπεθρο είναι μια αντικειμενική διαδικασία. Οι διαρθρωτικές αλλαγές γίνονται και θα γίνονται. αλλάζουν οι θέσεις απασχόλησης, δημιουργούνται, χάνονται. Το θέμα είναι οι υπηρεσίε που προσφέρουν οι γεωργοί. Μερικέ φορέ είναι αυτοαπασχολούμενοι, άλλε φορέ έχουν άλλου εργαζόμενου. Επίση, το θέμα τη παροχή υπηρεσιών, όχι μόνο για του ε, γεωργού που απασχολούνται, αλλά και για του κατοίκου ε, τη ε, υπαίθρου. Και το θέμα της τιμής των αγροτεμαχίων επίσης είναι σημαντικό θέμα. Ε, πάντως η ύπεθρος είναι πολυλειτουργική θα πρέπει να την ενισχύσουμε και επίσης υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα μέτρο για να το εφαρμόσουμε σε όλες τις χώρες. Είναι μεγάλες οι διαφορές μεταξύ τους. Και τέλος, ε, αν θα πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί δεν είναι επιβεβαιωμένη αυτή η πληροφορία, αλλά ακούσαμε Ακούμε που και που ότι τα προβλήματα της ανάπτυξης της υπαίθρου θα πρέπει να περάσουν από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που είναι πολύ σημαντικό για την κοινή γεωργική πολιτική να περάσουν από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, ε, Συνοχής Αυτό το αναφέρει και το σχέδιο του Γιούνκερ. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση. Δεν μιλάω για το στρατηγικό σχέδιο, αλλά για τη νέα προσέγγιση της κατανομής των δραστηριοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε βέβαια και ίσως να θέσουμε και σχετικές ερωτήσεις στον αρμόδιο επίτροπο, αλλά και στον πρόεδρο Γιούνκερ, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν επιβεβαιωθεί αυτή η μετάβαση ή η η αρμοδιοτήτων, και το διεθνές εμπόριο περάσει από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη στη Γενική Διεύθυνση Trade, φαντάζομαι αυτό που θα μείνει στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη είναι μια πολύ, ένα πολύ συγκεκ... συρρυκνωμένο πεδίο αρμοδιοτήτων και κυρίως και είναι η ορική πολιτική. Αυτή η συρρήκνωση των αρμοδιότητων τη Άγκρη είναι πολύ σοβαρό. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτέ οι πληροφορίε. Φημολογούνται όλα αυτά, αλλά ακούγονται αριστερά και δεξιά. Πάντω όταν επιβεβαιωθούν και επισημοποιηθούν αυτέ οι πληροφορίε, μάλλον θα είναι αργά. Θα βρεθούμε πρωτοτελεσμένο γεγονότο. Οπότε συμπαθάτε με που έθεσε το ζήτημα τώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό και ακόμη και αν δεν είναι επιβεβαιωμένε αυτέ οι πληροφορίε, νομίζω ότι ήταν σωστό να το θίξουμε. Κλείνω με αυτό το σημείο. Ευχαριστώ του ε, εμπειρογνώμονε γιατί και το θέμα ήταν σημαντικό και η συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Ε, πρέπει να γίνει αλλαγή εδώ των εμπειρογνωμόνων. Πολύ σημαντικό το θέμα και γι' αυτό θα ήθελα και ησυχία στην αίθουσα. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 13 που προβλέπει η ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα εργασίας για τις γεωργικές αγορές. Η ομάδα αυτή συγκροτήθηκε από τον αρμόδιο επίτροπο για να εξετάσει την κατάσταση στις γεωργικές αγορές. Επίσης, εξετάζει τη μεγάλη σημαντική επιρροή των εξωτερικών παραγόντων στην γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύει λοιπόν την κατάσταση των γεωργικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολείται με θέματα όπως η διαφάνεια της αγοράς, η πρόσβαση των γεωργών σε χρηματοοικονομικά μέσα, προθεσμιακές αγορές. Πολύ σημαντική αυτή η ομάδα εργασίας λοιπόν. Απαρτίζεται από 12 μέλη και παρακαλώ τους εκπροσώπους τους ε, να λάβουν θέση στο βήμα. Ο Επίτροπος Χόγκαν πολύ συχνά αναφέρθηκε σε αυτή την ομάδα εργασία ε, για τις διορικές αγορές με πρόεδρο τον κύριο Βέρμαν. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τη συζήτηση. Μας ενδιαφέρουν ε, οι εργασίες σας ε, και οι προτάσεις για το πώς θα διέλθουμε από την κρίση στη Γεωργία. Επαναλαμβάνω, είναι 12 μελής αυτή η ομάδα εργασίας, η Task Force. Θα σας δώσω 10 λεπτά, κύριε Βέρμαν. Μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Και κατόπιν στα μέλη της Επιτροπής σας που ήρθα μαζί σας και στους συναδέλφους στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό κύριε Βέρμαν σας παρακαλώ λάβετε το λόγο. This one, yes. Oh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά έρχομαι εδώ σήμερα. Να εξηγήσω τι κάνει αυτή η Task Force. Αυτή η ομάδα εργασία και τα καθήκοντα που καλούμαστε να επιτελέσουμε. Το καθήκον λοιπόν ξεκάθαρο, το όρισε ο Επίτροπος Χόγκαν, και αφορά την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην διτροφική αλυσίδα που έχει μεγάλη σημασία σε έναν κόσμο με περισσότερο ανθρώπους προς αγορές και παγκοσμιοποίηση ως προς τη διτροφική αλυσίδα. Τρο, ε, πρόθεσή μας αλλά και καθήκον μας δεν ήταν να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αναθεώρηση της ΚΑΠ. Θα ήταν υπερβολική με τα διαπέτηση για μια ομάδα Απλώς θέλουμε να βελτίωσουμε τη θέση του Γεωργού στη διατροφική αλυσίδα. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, με τι μέσα, τι στοιχεία υπάρχουν για την υλοποίηση του στόχου. Η ομάδα εργασία απαρτίζεται από πυρογνωμόνε των κρατών μελών που έχουν επιλεγεί επί τη βάση μια προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στην ομάδα εργασία με βάση την οποία προχώρησε σε επιλογέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογα με τη χώρα, το φύλλο, την πραγματογνωμοσύνη που διαθέτει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις υπηρεσίες της. Έγιναν, ε, έγινε μία από τις επτά σχεδιασμένες ε, συνεδριάσεις. Έχουμε προβλέψει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να είναι έτοιμη η έκθεση και πάντως πριν από το τέλος του 2016. Μας πιέσει ο Επίτροπος Χόγκαν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην ξεπεράσουμε το πρώτο του 2016. Με την έκθεση τρεις συνεδριάσεις μέχρι τώρα. Πολλά τα θέματα, θα τα καταθέσω σαφέ και για σας, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να σας τα ονόματα των ειδικών μας, των εμπειρογνωμόνων, μελών της Επιτροπής μας και της χώρας τους. From την Πολωνία εμπειρογνώμονα σε θέματα τροφίμων και παραγωγής τροφίμων. Κασολάρι from Italy. Από την Ιταλία. Ειδικό σε συνεταιρισμούς. The UK. Τον κύριο Τόπιν από το Ρωμανό Βασίλειο. Γαλακομικά. Fresco from the Netherlands. Κάτω χώρες. Πανεπιστήμιο. Βάχενιγκεν. Πρίτανης και ειδική βέβαια στη, στο τρόφιμο και τη Γεωργία, ο κύριο Γκίσεν της Γερμανίας, από τη Westflash, πρώην ε, Γενικός Διευθυντής και ο κύριος δίπλα μου, Βάρσον, που είναι ειδικό στις αγορές των παραγωγών, η κυρία Ιούας από την Ουγγαρία, Διευθύντρια Ερευνητικού Κέντρου Γεωργίας της Ουγγαρίας, κυρία Μπομιέ, Γαλλία αγορές παραγόγων στην ε, Γαλλία Μπεντζιέ πάλι εδώ στα αριστερά μου αναπληρωτή γενικός διευθυντής της Καρφούρ της Γαλλίας και η κυρία Βαλβέρντε Καβρέρο από την Ισπανία, Γενική Διευθύντρια σε Υπουργείο της Ισπανίας και ο κύριος Σαμίρ από τη Σλοβακία γνωστό, γνώριμο σας εδώ στις Βρυξέλλες, αφού είχε συμμετάσχει στις συνομιλίες και τις πραγματεύσεις για την προσχώρηση της Σλοβακίας στην Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η ομάδα εργασίας. Με χαρά σημειώνουμε ενεργό συμμετοχή από διάφορες χώρες, για διάφορες πτυχές, με διάφορους τομείς γνωστικούς και Τώρα, πέραν διαφόρων ζητημάτων ε, που έχουμε να ετοιμάσουμε, θέλουμε και να ξεκαθαρίσουμε λίγο την εικόνα και να προσκαλέσουμε ε, πράγματα γνώμονες από διάφορους τομείς ειδικού. Με πρώτο θέμα τη διαφάνεια των αγορών και τα δεδομένα τα σχετικά με τις αγορές. Πώς δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των αγορών έτσι ώστε ο παραγωγός να έχει στη διάθεσή του αξιόπιστα στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για σχεδιασμό, για λήψη αποφάσεων, να αγοράσει, να πουλήσει, να οργώσει, να σπείρει, να αρμέξει και ούτω καθεξής. Δηλαδή για να κάνει καλά τη δουλειά του και να κερδίζει ένα καλό εισόδημα. Διαφάνεια στην αγορά λοιπόν. Πολύ σημαντικό. Οι δύο εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένας και οι δύο άλλοι, σύνολο δύο, από τις πολιτείες, μας έδωσαν στοιχεία για την ε, διαφάνεια της αγοράς και για συστήματα και διαδικασίες που θα επιτρέπουν και πιο πρόσφατα αλλά και πιο αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες για την ε, τιμή που αντέχουν οι αγορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και τις προοπτικές είτε σπάνιδος, είτε ε, πληθώρας τροφίμων, συγκεκριμένων τροφίμων. Τα παράγωγα μετά. Παράγωγα και αγορές παραγόγων. Και εδώ μας απασχολεί το εάν είναι δυνατόν, αν είναι χρήσιμο, να χρησιμοποιηθούν προθεσμιακές αγορές για να ελέγξουν να συγκρατήσουν διακυμάνσεις τιμές που μπορεί να είναι και πολύ σοβαρές μάλιστα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο σε ένα κόσμο που η ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια κυρίως έχει ανοίξει τη σιγορά της έχει καταργήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις και τους μηχανισμούς ανθρωπίσης. Είναι πιο πληκτικές λοιπόν οι τιμές όπως δημορφώνονται, δεδομένο πια καθημερινό για τον Γεωργό και πρέπει να δούμε εάν οι προθεσμιακές αυτές αγορές μπορούν να χρησιμεύσουν για την ε, υποβάθμιση και διάδοση ταυτόχρονα του κινδύνου για το γεωργό και βέβαια το καταναλωτή. σε σχέση με το ποιος θα παραγάγει και ποιος θα πουλήσει το προϊόν. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Θα σας μας βοηθήσει όμως ο συνάδελφος που είναι ειδικό στο θέμα αυτό. και θα μας μιλήσει για το συγκεκριμένο αυτό το εργαλείο. Τρίτο θέμα, οι συμβάσεις και πώς αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερά εισοδήματα και να αντιμετωπίσουν την δυτικότητα των αγορών και τις εξελίξεις. Η συμβάση βέβαια είναι γνωστή λύση. Κοιτάμε όμως πώς μπορούμε να αναπτύξουμε με τρόπο πιο ομοιογενή, πιο ομοιόμορφο και πιο συμβατό αλλά και διαφανή τις συμβάσεις αυτές. Επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, έχουμε οικονομικές ενισχύσεις από διάφορα ταμεία, το περίφημο Ταμείο Γιούνκερ βέβαια, για την υποστήριξη της καινοτομία στο γεωρικό τομέα και τις εξελίξεις στην Ήπεθρο, προκειμένου να στηριχθούν οι γεωργοί σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Στόχος της μελέτης είναι περισσότερο να ακούσουμε από εσά τα σχόλιά σας και να πάρουμε από εσά ιδέες, τι ζητάτε ακριβώς. Έχουμε ιστότοπο στον οποίο περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις και τις ιδέες σας, θα τις λάβουμε υπόψη οπωσδήποτε. Και έτσι, κύριε Πρόεδρε, Είμαστε όλο αυτιά. Και σας βεβαιώ πως οι προτάσεις, οι ιδέες, οι συστάσεις σας θα σταθμιστούν και θα εξεταστούν με μεγάλη προσοχή μέσα στην Task Force. Σας ευχαριστώ. Ε, Φαντάζομαι η τα μέλη της ε, ομάδας εργασίας που σας συνοδεύουν θα δώσουν απαντήσεις και θα σχολιάσουν αυτά που θα ρωτήσουν οι ευρωβουλευτές. Ναι, όντως κύριε Πρόεδρε. Και είναι πρόσδεκτα όλα τα σχόλια της Επιτροπής σας. Όπως είπα, είμαστε αλευτιά. Θέλουμε να ακούσουμε από εσά τι σχόλια έχετε τις, ε, και τι ιδέες έχετε, πώς να ενισχύσουμε τη θέση του Γεωργού στην επιστηστική αλυσίδα. Δώστε μας προτάσεις, παρατηρήσεις, θα τα σημειώσουμε όλα αυτά προσεκτικά και θα τα εξετάσουμε επισταμένως. Η κυρία Αγγιλέρα, εκ μέρους των Σύλλης Δημοκρατών. Δύο λεπτά παρακαλώ κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε εμπειρογνώμονε της ε, Task Force αυτής της ομάδας εργασίας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα της ε, ανάλυσης ε, με τους εμπειρογνώμονες την κατάσταση αυτή που είναι μια κατάσταση μόνιμης κρίσης και αβάσταχτης για πολλούς επιμέρους κλάδους της γεωργίας. Έχουμε μια κατάσταση στην επιστημιστική αλυσίδα όπου φέρνει τον Γεωργό να είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Έχουμε απότομες διακοιμάσεις, μεγάλη αστάθεια των τιμών ε, που θίγουν κυρίως τους γεωργούς, ε, που είναι και στην πιο αδύναμη θέση. Θα πρέπει όλα αυτά να τα αναλύσουμε και να κάνουμε μια σωστή διάγνωση πριν προτείνουμε λύσεις. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους μηχανισμούς ρύθμισης των αγορών. Δεν έγιναν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ή προσαρμογές για τους μηχανισμούς διαχείρισης των κρίσεων, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την κρίση. Εγώ δεν πιστεύω στο αποθεματικό της κρίσης. Δεν πιστεύω σε ένα σύστημα που βγάζουμε από τον πρώτο πυλώνα χρήματα για να τα μοιράσουμε στους γεωργούς όταν διανύουν κρίση. Ή να πρέπει οι ίδιοι γεωργοί από μόνοι τους να λύσουν μια κρίση που δεν την προκάλεσαν γιατί είναι πολιτικού χαρακτήρα ή άλλου τύπου. Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει η κοινωνική πολιτική με τη μεταρρύθμιση. Με τα εργαλεία που έχουμε και τους μηχανισμούς, αναφερθήκατε σε κάτι στη μελέτη σας που είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε την κατάσταση της συμβάσης, να δούμε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις στη Γεωργία. Εγώ είμαι Ισπανίδα και στη χώρα μου Έχουμε συμβάσεις, υποχρεωτικές μάλιστα συμβάσεις, ε, μονοετής, ε, στο γαλακτοκομικό τομέα και παρόλα αυτό ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα. Οπότε με ενδιαφέρει ιδιαίτερος ε, να βρούμε τρόπο για να εξασφαλίσουμε μέσω των συμβάσεων τα γεωργικά εισοδήματα. Γιατί μέχρι στιγμής έχω πολλές αμφιβολίες για το αν εφαρμόζονται σωστά οι συμβάσει. Πιστεύω επίσης στη διαφάνεια της αγοράς. Θα πρέπει τα στοιχεία να γνωστοποιούνται. Και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως τα αποτελέσματα ε, τη εφαρμογή των προθεσμιακών αγορών για μερικούς τομείς. Ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία γιατί ε, από τα δικά σας θετικά αποτελέσματα θα εξαρτηθεί και βελτίωση κατάσταση στη Γεωργία. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστούμε κύριε Βέρμαν. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Είστε ευπρόσδεκτοι στην Επιτροπή μας. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπατε. Και ε, συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας με ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολύ αντίξωες ηθίκες και ίσως σε μία από τις χειρότερες κρίσεις που αντιμετωπίζει η Γεωργία στην Ευρώπη. Γιατί σε μεγάλο βαθμό ε, είχαμε ε, το ρωσικό εμπάργο, την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, την πτώση των τιμών, τη θέση της Κίνας, ε, το ιστορικό υπόβεθρο του το γνωρίζουμε. Σας ευχόμαστε καλή τύχη, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο σας και πολύ περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα πορίσματα της έκθεσής σας. Ελπίζω όντως να εκφωνήσετε την έκθεσή σας το συντομότερο δυνατό και ελπίζω να μην έχει την ίδια μοίρα που είχαν άλλες εκθέσεις στο παρελθόν. Δηλαδή να μπουν στο χρονοδούλαπο και να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Θέλουμε να αξιοποιηθεί η έκθεσή σας και να φέρει θετικά αποτελέσματα. Αναφερθήκατε σε κάποια προβλήματα της επισητιστικής αλυσίδας. Φαντάζομαι στην έκθεσή σας θα ασχοληθείτε και με θέματα όπως οι προθεσμιακές αγορές, οι νέες αγορές, οι νέες διέξοδοι, οι νέες ιδέες, οι νέες προτάσεις. Πόσα θα διαθέσουμε τα προϊόντα μας. Και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, το γνωρίζετε. Υπάρχει μεγάλη δυσπιστία μεταξύ του παραγωγού και του μεταποιητή. Δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών. Και γι' αυτό είναι πολύ ζωφερό το μέλλον στο γαλακτοκομικό τομέα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε καλύτερη συνεργασία. Είπατε συμβάσει. Ίσως είναι μια καλή λύση. Αλλά ε, στις προθεσμιακές αγορές εκεί και αν υπάρχει δυσπιστία και καχυποψία. Γιατί όλοι μας λένε καινούριο είναι αυτό το θέμα, πρώτη φορά το βλέπουμε. Πώς θα το προβάλλουμε λοιπόν στον κόσμο για να τους προσελκύσουμε. Γιατί και μένα με ρώτησαν και εγώ όπως και εσείς περιμένω και τις προτάσεις των άλλων και τα σχόλια των άλλων και τις κρίσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχει λειτουργήσει το NMO. Πάντως αυτό που πρέπει να κάνουμε και το πιστεύω ειλικρινά είναι ότι δεν θα πρέπει να καθόμαστε με, τα, με σταυρωμένα χέρια και να περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νέα Ζηλανδία ή οποιοδήποτε άλλον να θέσουν τις αρχές, τις προδιαγραφές ε, για τις τιμές των ε, γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα πρέπει εμείς να πρωτοστατήσουμε, εμείς να είμαστε πρόδρομοι και να υποβάλουμε προτάσεις για να προστατεύσουμε το γαλακτοκομικό μας τομέα, να θέσουμε τις αρχές, τα επίπεδα και τις προδιαγραφές δεν αρκεί το παρατηρητήριο για το γάλα που έχουμε. Χρειάζουμε, ε, χρειαζόμαστε δίκαιη τιμή όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και μια αξιοπρεπή τιμή για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Κύριος Χαϊτεμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε κύριε Φρέμα που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μα για να μα μιλήσετε για αυτήν την ομάδα δράση. Για να είμαι ειλικρινή, πραγματικά χαίρομαι που υπάρχει μια τέτοια ομάδα δράση για τι γεωργικέ αγορέ. Το βρίσκω πολύ σημαντικό. Αλλά έχω μια ερώτηση για εσά. Τι πιστεύετε ως πρόεδρος για τη δουλειά της ε, Task Force, πιστεύετε ότι είναι επιτυχημένη. Σημαντικό είναι να βγει κανείς και λίγο από το ρόλο του για να δει τα πράγματα απ' έξω. Επίσης, για ένα από τα ζητήματα που θίξατε, τη διαφάνεια των αγορών, τα ασφαλιστικά συστήματα και τα χρηματοδοτικά συστήματα. Για τη διαφάνεια της αγοράς, βλέπετε ίσω και τι αρνητικέ συνέπειε μπορεί να έχει, πώς μπορεί να γυρίσει ως μπούμερανγκ για του γεωργού, ότι οι λιανοπολιτέ μπορούν να την ε, χρησιμοποιήσουν καταχρηστικά για να πιέσουν προ τα κάτω τις τιμέ των γεωργών. Και ω προ τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τι ασφαλίσει αυτό δεν είναι καινούριο. Κάποιοι τομεί ανατρέχουν σε αυτά περισσότερο από ό,τι άλλοι, κάποια κρατημέλη επίση, αλλά λόγω χάρη ο νόμο περί τον είπα, έχει πολύ συγκεκριμένε διατάξει για τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα κοιτάτε αυτά και κάνετε τι απαραίτητε συγκρίσει. Και ακόμη πιο ε, συγκεκριμένα για τα ασφαλιστικά προγράμματα και τι ασφαλιστικέ διατάξει. Κατά την άποψή μου, αυτό που θα βοηθήσει του γεωργού να αντιμετωπίσουν προληπτικά του κινδύνου και να στραφούν με καλύτερο τρόπο προ την αγορά, αλλά ίσω και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά, είναι ακριβώ αυτά τα συστήματα. Το πιστεύετε αυτό, ή πρέπει να είναι ανεξάρτητη η στήριξη του εισοδήματο των γεωργών. Πάντως, προς στιγμήν υπάρχουν κάποια ασφαλιστικά προγράμματα που ήδη ε, ισχύουν, όπως μπορεί κανείς να ασφαλιστεί λόγω χάρη για κακές μετεωρολογικές συνθήκες. Όμως αυτά τα ε, ασφαλιστικά συστήματα δεν τα αξιοποιούν αρκετά ακόμα οι Γεωργοί. Γνωρίζετε γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί λόγω χάρη οι Γεωργοί δεν αυτοδιοργανώνονται σε οργανώσεις παραγωγών ή έστω σε συνεταιριστικέ οργανώσεις. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που του εμποδίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σέντρα. Σέντρα. Κυρία Σέντρα. Σέντρα. Ε, Ευχαριστώ. Δεν είχα ζητήσει το λόγο νομίζω κύριε Πρόεδρε, αλλά μια και μου τον δίνετε θα τον χρησιμοποιήσω. Μα ήθιστε να δίνω το λόγο συστηματικά στους συντονιστές, γι' αυτό σας τον δίνω. Α, καλώς, εντάξει, ευχαριστώ, τίποτα, εντάξει. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα συνεχώς. Και όταν μιλούμε για τις γερικές αγορές, έχω την αίσθηση ότι όλες οι συζητήσεις που γίνονται εστιάζονται πάντα στο ίδιο θέμα, στις αγορές εξαγωγών και το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε στο γαλακτοκομικό τομέα μιλούμε μήνες ολόκληρους για αυτό το πρόβλημα και σε άλλους γεωργικούς τομείς το πρόβλημα είναι ότι αναζητούμε συνεχώς μηχανισμούς για να βρούμε εμβαλωματικές λύσεις σε αυτή την απορρίθμιση που προκάλεσε μία μικρή ομάδα που προσανατολίζεται προς τη διεθνή αγορά. Ερωτώ λοιπόν, πότε επιτέλους ε, θα ασχοληθούμε και ε, οι εμπειρογνώμονε και αυτή η ομάδα εργασία και τι γεωργικέ αγορέ για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίε γεωργικέ εκμεταλλεύσει, που με την πολιτική μας ε, για τις εσωτερικές αγορά συνεχώ του οδηγούμε, του τριμώχνουμε στον τοίχο, του οδηγούμε στην πτώχευση ή στην μόνιμη κρίση. Μα μιλήσατε για διαφάνεια των αγορών, μα μιλήσατε για ασφαλίσει, προθεσμιακέ αγορέ. Εντάξει, μία από τα ίδια, αλλά η κρίση συνεχίζεται. Επιτέλους, ας ασχοληθούμε με την πραγματικότητα, με τους χωρικούς, με τους αγρότες και τις αγρότητες, του πραγματικού κόσμου και όχι ε, για αυτές τις μικρές ομάδες, τις ολιγομελείς ομάδες που επιζητούν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Κύριε Χόισλινγκ, σας ενδιαφέρει ο λόγος. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι μια κάποια απογοήτευση. Βλέποντας εδώ την επιτροπή αυτή που μας παρουσίασε. Εκπρόσωπος της Γεωργίας προβλέπετε. Α, καλά, ναι. Ένας από τους 12. Μα είναι κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Η Best flies της Γερμανίας. Μαζί με τον μικρό παραγωγό είναι δυνατόν να μιλάει για διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι ακριβώς όπως σας το περιγράφω. Γιατί να μην υπάρχει κανεί ο οποίος να εκπροσωπεί, βγάλετε τον αυτό από την υπόθεση, από καταμέτρηση, να εκπροσωπεί τη γεωργία, τον μικρό παραγωγό. Μιλάμε για διαφάνεια. Με τουλάχιστον 50 εκθέσεις τα τελευταία 5 χρόνια εκπονήσει στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό ακριβώς, για την έλλειψη συμμετοχής του γεωργού στην ε, αλυσίδα της ε, ε, διάθεσης στην αγορά των προϊόντων. Στάχτη στα μάτια είναι αυτά που μας λέτε εδώ. Μιλάτε για ε, προθεσμιακές αγορές, για μεταρρυθμίσεις. Μα τα έχουμε συστήσει όλα αυτά με την ΚΑΠ. Κάθε δυνατή λύση για τη γεωργία την έχουμε συστήσει εδώ. Εάν αυτό που μας προτείνετε ως λύση είναι αυτό εδώ που μας δείξατε, αυτή η σύνθεση, τότε δεν βλέπω κανένα μέλλον. Κοιτάξτε λίγο τι δικέ μα εκθέσει αυτά που έχουμε εμεί ετοιμάσει ω Κοινοβούλιο, γιατί μπορεί να σα δώσουν και κάποιε ιδέε για απάντηση. Μπορεί να σα φανούν και χρήσιμα. Το δικαίωμα στον ανταγωνισμό πρώτα απ' όλα. Είναι άδικο το δίκαιο του ανταγωνισμού στη, στον τομέα τη γεωργία. Το καρτέλ πρέπει να τα συζητήσουμε. Πού είναι τα δικαιώματα των παραγωγών στην αλυσίδα. Πρέπει να τους ενισχύσουμε και δεν άκουσα την αρέτη κουβέντα ούτε εσείς. Μιλήσατε για προθεσμιακές αγορές. The American way of agriculture. Όπως κάνουν οι Αμερικάνοι δηλαδή. Μα δεν γίνεται αυτό. Έγινε χθες ενδιαφέρουσα συζήτηση. όπου ακούστηκε και το ενδεχομένως ε, ε, να έχουμε εμείς ε, κάνει το λάθος να μειώσουμε το συμφέρον μας, να πλήξουμε τα ίδια μας τα συμφέροντα με την κατάργηση των κοινών οργανώσεων, με την εξέλιξη των κοινών οργανώσεων αγοράς. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε και έτσι όπως θα παρουσιάζετε εσείς τον ε, παραγωγό δεν θα τον βοηθήσουμε. Δεν δεν έχουμε γεωργούς ε, στην αίθουσα γιατί ήρθε η Άνοιξη και οι γεωργοί είναι στα χωράφια τους. Ο κύριος Άγνιο. Μα δεν είχα σηκώσει την κάρτα μου γιατί δεν ήξερα αν θα μπορούσα να μείνω μέχρι το τέλος της συζήτησης. Χαίρομαι που έμεινα όμως. Μιλήσατε για τις προθεσμιακές αγορές. Εγώ προσωπικώς τις έχω αξιοποιήσει, είναι χρήσιμες, αποδεδειγμένα. Αλλά φαντάζομαι και να έχετε υπόψη ότι σε αυτό το θεσμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει νομοθεσία MIFID, η οποία θα καταστήσει πιο δύσκολη την ε, ε, χρήση των προθεσμιακών αγορών. Δεν ξέρω γιατί θέλω να το κάνω αυτό, μην μου φαίνεται το παραγωγικό. Φαίνεται να θεωρούν ότι οι αγορές προθεσμιακές αναεβάζουν την τιμή των τροφίμων. Ε, για μένα καθόλου ε, δεν είναι σωστό αυτό. Αντιθέτως, μπορούν να αποστείλουν πολύ χρήσιμα μηνύματα στις κυβερνήσεις και του καταναλωτές και του παραγωγούς. Θα υπάρξει νέο δημοψήφισμα, όπως ξέρετε, τις επόμενες εβδομάδες στην πατρίδα μου. Ο νέο υπουργό Γεωργίας Τίζεται υπέρ του... Ε, ναι, υπέρ του να αποχωρήσει δηλαδή η Βρετανία από, το, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συστήματα λοιπόν προσδιορισμού τιμών που έχει εισαγάγει και ο Καναδάς και τα οποία υποστηρίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι εξασφαλίζουν σταθερότητα. Ο κάθε καταναλωτή η κάθε διαδικασία παραγωγή γεωργικών προϊόντων χρειάζεται μία εγγυημένη βάση προμήθειας των προϊόντων. Δεν μπορεί να λέει θέλω το ίδιο προϊόν για λιγότερα χρήματα του χρόνου. Γιατί είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ε, κατακόρφη ολοκλήρωση βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε ό,τι μα έρχεται και μετά να λέμε στον πολιτικό «Για σε παρακαλώ να μου βρει έναν τρόπο να διαθέσω το προϊόν μου κερδίζοντας και εξασφαλίζοντας και κέρδος». Η κατακόρυφη αυτή λοιπόν ολοκλήρωση σημαίνει ότι η διαδικασία από την παραγωγή, την προμήθεια ε, και μέχρι την κατανάλωση πρέπει να ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους ε, τομείς, ε, κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να περνάει από τη δικασία την ασφαλιστική, να φτάνει μέχρι το σούπερ μάρκετ που θα πωλεί τελικά το προϊόν στον καταναλωτή, με ένα προϊόν το οποίο θα ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα ξέρει ο καταναλωτής όταν το αγοράζει ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον της γεωργίας στα τρόφιμα. Κυρία που είναι η συγγήτρια για το θέμα της επιστηστικής αλυσίδας. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ήταν σοφή η παρουσίασή σα. Με ενδιέφερε μετά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στι 13 Ιανουαρίου και πολύ εντατική εδώ για την αγορά που καθορίζει μόνο τις τιμέ. Το θέμα είναι οι φορεί τη αγορά, πώ λειτουργούν, γιατί δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι η αγορά μόνο της καθορίζει τις τιμές και τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζουν. Βλέπω εδώ στο κείμενο το εδάφιο που λέτε ότι πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν στις εθνικές ρυθμιστικές προσπάθειες και την ε, προσπάθεια των κρατών να ελέγξουν τις εμπορικές πρακτικές και την ε, ε, διαμόρφωση των τιμών. Και υπήρξε έκφραση αμφιβολιών. Εδώ υπάρχει μια συνέπεια, διότι οι αθέμητε εμπορικέ πολιτικέ δεν έπρεπε να υπάρχουν καν. Και ό,τι χρειάζεται για να εκριζωθούν πρέπει να γίνει. Αυτό πιστεύει αυτή η Επιτροπή, ότι χρειάζεται τέτοιου είδους ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι πρέπει να πείσουμε τους πάντες να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η έννοια της ενίσχυσης της θέσης των ε, γεωργών ποτέ δεν ακολουθείται από την άλλη ιδέα. Γιατί επιτρέψαμε στους άλλους να πάρουν τέτοια δύναμη. Ίσως λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα πάρουμε τη δύναμη από αυτούς που έχουν πάρα πολύ ε, μεγάλη εξουσία στα χέρια τους στην ε, αλυσίδα παροχής τροφίμων, την αλυσίδα πώληση των τροφίμων. Πρέπει να δούμε πώς ένας επιχειρηματίας μπορεί να πάρει την εξουσία από τα χέρια ενός μικρού γεωργού που παράγει. Επίσης, για τους καταναλωτές και την προστασία τους και τη διαφάνεια. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια τιμών για τους καταναλωτές. Δηλαδή, όταν πάνε σε ένα λιανοπολίτη για να ψωνίσουν κάτι, αυτό που βλέπουν στην ετικέτα δεν είναι όλη η αλήθεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια σαφή διαδικασία για τον υπολογισμό του κόστους και της ωφελίας. Κυρία Χάζεκαμπ, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε κύριε Βέρμαν. Όπως θα φαντάζεστε, θα σας μιλήσω για εντατική κτηνοτροφία. Λίγοι το τομεί. που χτυπήθηκαν τόσο πολύ για τόσο καιρό από την κρίση. Οι τράπεζες είναι ένας τομέας, τραπεζικός τομέας, όπου τα πράγματα πήγαν από το κακό στο χειρότερο και η Γεωργία επίσης. Απότομες διακοιμάσεις τιμών και αύξηση παραγωγής που δεν βοήθησε φυσικά τη σταθεροποίηση των τιμών ή την αύξησή τους. Το διαπιστώσαμε αυτό και στο βόλιο κρέας και στο γαλακτοκομικό τομέα. Υπάρχει κορεσμός. Και στο παρελθόν είχαμε ως στόχο την αύξηση της παραγωγής, αλλά στο μεταξύ το σύστημα πήγε κατά διαβόλου. Το 80% των ε, γεών και των ε, γεωργικών εκτάσεων ε, από το 50% ε, αφιερώνεται στην καλλιέργεια δημητριακών για την παραγωγή ζωοτροφών. Ε, εντατική κτηνοτροφία, επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, απερίμωση, λιμοκτονούν πολλές γεωργικές κοινότητες, εσείς ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας, τι λύση προτείνετε. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις για να τεθεί επιτέλους ένα τέρμα σε αυτή την εντατική κτηνοτροφία. Κυρία Σρέιερ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζονκαμπ. είπε μερικά πράγματα που τα βλέπω και εγώ στη χώρα μου, αλλά κύριε Βέρμαν, σας έχω ήδη δει ε, να δουλεύετε στην ε, γεωργία με τα ρούχα εργασίας. Τέλος πάντων, στις κάτω χώρες αυτό που λέμε είναι ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχει ήδη επηρεάσει πάρα πολύ το γεωργικό κλάδο. Το είπε και η κυρία Μαγκίνος. Το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα τα μπλοκάρουν οι διανομής. Δηλαδή, εάν δεν βρούμε μια συμφωνία με αυτού που διανέμουν τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στου ίδιου του γεωργού. Τι γνώμη έχετε εσεί. Έπειτα για το ε, ψηλότερο κόστος και την ε, καινοτομία στι αγορέ, Αυτό δεν είναι προνόμιο του μόνο των κάτω χωρών. Απλώς εσεί ήσασταν από του μεγάλου εμπνευστέ αυτή τη προσπάθεια. Πιστεύετε ότι η κατάσταση είναι ισότιμη στην Ευρώπη, διότι όταν έχει κανεί υψηλότερε απαιτήσει, δεν πρέπει να απαιτεί το ίδιο και από του ανταγωνιστέ του. Το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας έχει εξηγήσει ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις πρέπει να προστατεύονται. Αλλά θεωρεί καθοριστική σημασία και τον ανταγωνισμό. Να το θυμηθείτε κι εσείς και να το ε, αναφέρετε προ τα ασφαλιστικά ταμεία, ω προ το πρόγραμμα Juncker και του παραγωγού. Ωραίο εργαλείο είναι αυτό και το έχουμε συζητήσει πολύ, αλλά τι συμβαίνει στην πράξη. Οι γεωργοί δεν έχουν δικαίωμα να αυτοκαθορίζονται. Εσείς τι θέλετε να προωθήσετε, τους, τις πολυεθνικές, την υπερεπιδότηση ή τους μικρογεωργούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Φερμάν, ευχαριστώ για την ε, λευσή σας και τους συναδέλφους σας από την ομάδα δράσης. Εγώ είμαι υπεύθυνη για την έκθεση περί διακυμάτων τιμών. Υπό αυτήν την έννοια, πολλά ήδη υπόθηκαν βέβαια από του συναδέλφου, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει. Ε, μιλήσαμε για την ανταγωνισμό και τι αθέμητε πρακτικέ. Ε, εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τη διαφάνεια, γιατί την αναφέρατε. Ε, διερωτώ με, ως γεωργός η ίδια, γιατί είναι φορέα του αγροτικού κλάδου, λοιπόν. Τι εννοούμε με τη διαφάνεια. Τι θα πει διαφάνεια. Διαφάνεια θα πει ότι ο πρωταγωνιστής στην αγορά είναι ουσιαστικά ε, ικανός να σφετεριστεί, να εκμεταλλευτεί τον πιο αδύναμο. Μας ενδιαφέρει πώς θα προστατεύσουμε λοιπόν τα εισοδήματα των μικρών γεωργών. Διότι όταν μιλάμε για την διακύμανση των τιμών, εκείνοι είναι αυτοί που πλήττονται κυρίω. Ποια είναι η άποψή σα λοιπόν για το παρατηρητήριο των τιμών για, το, για τα αντασφαλιστικά ταμεία και για το τι μπορούμε να κάνουμε βλέποντας τα καλά παραδείγματα από άλλε περιοχέ του κόσμου. Θα είχα πολλές παρατηρήσει να κάνω δεδομένου του περιεχομένου τη εκθεσή μου, αλλά εφόσον χρειαστεί θα έρθω εγώ απευθείας σε επαφή με την δική σα ομάδα για να λάβω τις απαραίτητες απαντήσει. Βεβαίω, μπορείτε να στείλετε και γραπτό στις ερωτήσει σας στην ομάδα εργασία. Του εμπειρογνώμονε. Ο κύριος Δαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που μας διαθέτετε το χρόνο σας. Σήμερα μιλούμε για κρίση και να ζητούμε εργαλεία αντιμετώπισης αυτής. Για να μην πω θεραπείες. Είναι περιττό να θυμίσω ότι πριν από τρία χρόνια, όταν ψηφίσαμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αυτή βασίστηκε στην αρχή ότι δεν θα υπήρχαν πλέον κρίσεις, ότι οι αγορές θα αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο και ότι κάπως κάποιες μικρές μικροπροσαρμογές χρειάζονται. αλλά μας διέψευσε η αλληλουχία των γεγονότων. Άρα, η ερώτηση που θα σας θέσω είναι κάπως διαβολική και γι' αυτό σας έχουμε κάθε τύχη για να βρείτε μια απάντηση. Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Το έχω αναφέρει πολλές φορές εδώ, στην Επιτροπή μας. Εδώ και 60 χρόνια το δίκαιο περί ανταγωνισμού στην Ευρώπη έχει οικοδομηθεί προς όφελος και προς το συμφέρον του καταναλωτού. Η πολιτική αυτή ήταν τελείως λογική σε έναν χώρο όπου υπήρχε ένα 3-4% ανεργία. Σήμερα δεν πρέπει να σκεφτούμε τι νόημα πρέπει να λάβει η πολιτική του ανταγωνισμού σε έναν χώρο όπου έχουμε 10% ανεργία. Σε ποιο βαθμό το δίκαιο θα λειτουργεί ε, κατά των συμφερόντων των εργαζομένων, προστατεύοντας πάντοτε το συμφέρον των καταναλωτών. Ευχαριστούμε κύριο Μπούντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε αναλογιστεί τη δυνατότητα σύστασης μηχανισμών επέμβασης όταν ε, υπάρχουν επικίνδυνες ε, επιβλαβείς συμπεριφορές στην αγορά. Στην αγορά το χειρίου κρέατος, για παραδείγματι. Ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές στην ε, ευρωπαϊκή αγορά, συγκρίσιμες μεταξύ των κρατών. Α, στη Ρουμανία, ωστόσο, επί ένα χρόνο είχαμε φτάσει στο 0,75 ευρώ, 75 λεπτά του ευρώ, πολύ κάτω δηλαδή από την μέση τιμή των ευρωπαϊκών αγορών. Χρειάζονται λοιπόν μηχανισμοί παρέμβασης στις αγορές και σταθεροποίηση τους. Αυτό κράτησε ένα χρόνο στη Γερμανία. Πουλούνταν το κρέας, δηλαδή το, το χοιρινό, ε, σε τιμή κάτω του μισού του κόστους. Επίσης, πρέπει να υπάρξει κάποιο ομοιόμορφη, σχεδιασμό τη σχεδιασμός Πρέπει βεβαίως να κοιτούμε ποια είναι η αλυσίδα της ζήτησης και της προσφοράς, τι ζητάει η αγορά για να σχεδιάσουμε τις γεωργικές πολιτικές, που είναι και άλλωστε και δουλειά της Επιτροπής. Χρειάζεται να υπάρχουν οι σωστές πολιτικές, ώστε να μπορεί ο ε, παραγωγός να σχεδιάζει την παραγωγή του. Ευχαριστώ πολύ. Χόιμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολούθησα και εγώ τη συζήτηση και όχι μόνο την παρουσίαση αλλά και τα άλλα σχόλια και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτή η task force πιο πολύ στρέφεται προς την ε, μεταποίηση στη γεωργία και όχι την παραγωγή. Και αυτές τις οπτικές γωνίες εκφράσει λέτε ότι πρέπει, να είναι τα, δεδομένα να είναι ομοιόμορφα και συμβατά. Δεν ξέρω όμως εάν θα πρέπει εγώ να έχω σύμβαση ε, ισοδύναμη, συμβατή και ανταλλάξιμη με, του μεταποιητή στον οποίο πολλώ τα προϊόντα μου. Ε, υπάρχει τώρα φαίνεται η ιδέα να θεσπιστεί μια, ένα παρατηρητήριο της αγοράς του γάλακτος, αντίστοιχα με αυτό που υπάρχει για το βόλιο κρέας. Πώς λοιπόν έχετε ε, τα στοιχεία αυτά, πώς συλλέγονται τα στοιχεία αυτά και πώς τα διέθετε στην Επιτροπή. Τα στέλνετε πάντα στην Επιτροπή, θα γίνεται το ίδιο τώρα ε, μετά το παρατηρητήριο του γάλακτος και για το παρατηρητήριο για το κρέας. Ε, και πώς θα γίνεται η αξιολόγηση, θα γίνεται αξιολόγηση κινδύνου, το ξέρουμε αυτό, αλλά το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Για το γάλα πάλι. Ξέραμε αυτό καταβολικά, ότι με το τέλος των ποσοστώσεων υπήρχε κίνδυνος, ας το πω έτσι, ε, κομψά. Ε, ήρθε μετά η κατάργηση των ποσοστώσεων, ήρθε η εισβολή, να το πω κομψά πάλι, από την εξωτερική αγορά, από την παγκόσμια αγορά και τρίτος παράγοντα επιβαρυντικός, το εμπάρκο της Ρωσίας. Αυτά πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς όταν βλέπει ότι υπάρχει αυτή η τάση. Κύριος Γιάρ. Μια ναι, συμπληρωματική ερώτηση έχω. Οι προθεσμιακές αγορές, οι χρηματιστήρια, ε, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν στο να ε, προσδιορίσουν οι αγορές προς τα που θα τίνουν για το μέλλον, για να είναι αυτό πιο, γαρό, ναι, ε, πιο ορατό. Πολύ καλά, αλλά πώς μπορείτε να προσδιορίσετε αυτές τις τάσεις ώστε να προστατεύσετε την αγορά από την κερδοσκοπία, γιατί η κερδοσκοπία στα τρόφιμα είναι καταστροφή, ιδιαίτερα για τον ε, παραγωγό ο οποίος ε, άγεται και φέρεται. Γιατί, πώς λοιπόν μπορούμε αυτές τις προθεσμιακές αγορές και τα χρηματιστήρια να τις, ε, κοιτάξουμε, να τις αξιοποιήσουμε ώστε να φέρουν θετικά αποτελέσματα και όχι αρνητικά. Και επίσης ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να είναι προσβάσιμο στο γεωργό χωρίς επιπλέον κίνδυνο. Εάν μπορεί δηλαδή η αλυσίδα της αγοράς, η τροφική αλυσίδα της αγοράς να το αξιοποιήσει, μπορεί και ο Γεωργός, Κύριο Ντόρφμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω ότι ε, θα συμφωνήσω με αυτούς ε, που λένε ότι θα είναι περιορισμένα τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας εργασίας. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι θα έχετε καλά αποτελέσματα, αλλά κύριε ε, Βέρμαν, θα πρότεινα να κοιτάξετε και τι τύχη θα έχουν ε, τα πορίσματα της μελέτης σας, να μην μπουν σε ένα σιρτάρι δηλαδή και λησμονηθούν. Ε, έχουμε 55 δισεκατομμύρια προπολογισμό για την ε, Γεωργία. Είπαμε, υπόθηκε από όλους τους αδέλφους ότι έχει αμυντικό σχεδιασμό. Δεν υπάρχει μια ε, αποφασιστική, ε, επιθετική θα έλεγα πολιτική γεωργική, μόνο σε ορισμένους τομείς όπως εκεί όπου μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση αγοράς και βλέπουμε ότι εκεί κρίση, παραδόξως πως, δεν έχει εμφανιστεί. Άρα έχουμε και καλά αποτελέσματα χάρη στους οργανώσεις αγορές, αγοράς. Ε, θεωρείτε λοιπόν ότι είναι καθήκον σας να εξετάσετε και τους μηχανισμούς που ισχύουν αυτή τη στιγμή και λειτουργούν, πώς έχουν επηρεάσει την αγορά και πώς μπορούν στο μέλλον να την επηρεάσουν και αν χρειάζεται να εισηγηθείτε την εισαγωγή πολιτικών διαχείρισης αγοράς. Κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ. Κύριε Βέρμαν, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Γεωργίας. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ομάδα εργασία ε, στην οποία προεδρεύεται, για τις γεωρικές αγορές. Έχουμε και το φόρο με ψηλό επίπεδο για την καλύτερη λειτουργία της επισητιστικής αλυσίδα. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο ε, φορέων και κυρίω για τη δική σα ομάδα εργασία. Τι γίνεται με το άρθρο 222 και τα καρτέλ στην κρίση, τι διδάγματα άντλησε η ομάδα εργασία σα από την εφαρμογή του άρθρου 222. Επίσης, η διαπραγματευτική θέση των ε, παραγωγών, των γεωργών. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις θέσεις και, και τις προτάσεις σας και ελπίζω να είναι σημαντικές και αρέσουν. Κυρία Μίλλερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Έχω και εγώ ερώτηση σε σχέση με τα τρόφιμα και την αλυσίδα τη διατροφική. Έχουμε στη Γερμανία μια υπουργική απόφαση με έγκριση Υπουργού της Οικονομίας που τάσσεται κατά τον καρτέλ για την αλυσίδα διατροφική, οι δύο μεγάλες ε, εταιρείες σούπερ μάρκετ που είχαν συμφωνήσει ε, μεταξύ τους για τη χείριση αγοράς. Ε, Τάχθηκε κατά αυτόν λοιπόν ο υπουργό. Και επίσης θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το γάλα, εάν θα συμμετάσχουν μεγάλοι παράγοντες του γαλακτοκομικού τομέα, γιατί οι ε, ε, μικρές επιχειρήσεις γαλακτοκομικές δεν φαίνεται να έχουν ενδιαφέρον συμμετοχή. Σε αυτά ερωτώ λοιπόν ε, τρίτον εάν θα υπάρχουν συνδεμένες πρημοδοτήσεις για τα 27 κράτη με μόνη τη Γερμανία που έχει αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις και πώς τάσεστε ως προς την προσέγγιση αυτή. Γράψαμε όμως ότι μόνο το 13% ε, του γεωργικού προπολογισμού μπορεί να δοθεί στην στήριξη της παραγωγής. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ακόμη και αν οι γεωργοί συγκεντρωθούν σε ομάδες και κοινέ οργανώσεις παραγωγών, θα υπάρχουν ακόμα τεράστιες πολυεθνικές, θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από ότι αυτές οι οργανώσεις. Να πω είπε η κυρία Μαγκίνες, δύο πράγματα που να γίνουν, όχι μόνο να διοργανωθούν οι γεωργοί, αλλά και να περιοριστεί το μέγεθος των εταιριών με τους οποίες έχουν να κάνουν οι Γεωργοί. Η Επιτροπή φαίνεται να ενδιαφέρεται πάρα πολύ να προωθεί, να διώκει μάλλον εταιρείες όπως η Ryanair, η Microsoft, η Google κατά καιρούς, αλλά δεν πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο και στη Γεωργία και κάτι στο τοπικό επίπεδο βλέπουμε τη συγχώνευση της Slaney Foods και της EBP 40% του πρόβειου κρέατος στην Ιρλανδία. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Με τέτοιες καταστάσεις πάντοτε θα συγχλίβονται οι γεωργοί εκτός αν δημιουργήσουν τεράστιες οργανώσεις. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουν όμως και να πετύχουμε εμεί κάτι είναι να περιορίσουμε το μέγεθο αυτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι καταστάσει είναι ακραίε σε κάποιε ε, και χώρε. Υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα μαγαζιά και καταστήματα εδώ στι Βρυξέλλε, όσο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν ακόμη πολλά καταστήματα τροφίμων, πολλά ντέλη καταστήματα όπω λέγονται. Όμω όταν ε, τα μαγαζιά είναι στα χέρια μια εταιρεία, αυτοί αποφασίζουν τι γίνεται και αποφασίζουν σε, σε, όλη την, ε, σε όλο το μήκο τη αλυσίδα. Τι θα κάνετε λοιπόν για τον περιορισμό του μεγέθου των πολυεθνικών, διότι στο τέλο δεν θα προστατεύουμε του καταναλωτέ. Στο τέλο θα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θα έχουν την εξουσία στα χέρια του και θα του ε, τσακίζουν όλου. Κύριε Σροπέ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ασχολούμαστε με ένα πολύ σημαντικό θέμα και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Έχω και εγώ μερικές ιδέες. Όταν μιλούμε για διαφάνεια των αγορών, όσο και να μιλούμε για το θέμα αυτό, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση μόνο με τα λόγια. Αν δεν θεσπίσουμε ρυθμίσεις, τότε δεν πρόκειται να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια της αγοράς. Αν θέλουμε πραγματικά διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπίσουμε ελέγχους και κάποια στοιχεία εποπτείας της αγοράς. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Σας ερωτώ λοιπόν, τι γνώμη έχετε για την υποχρεωτική σήμαση, την υποχρεωτική ετικεταθεσία. Μόνο έτσι ο καταναλωτής ε, θα γνωρίζει πώς ο, τι, τι, τι με το λαμβάνει ο παραγωγός, ο μεσάζων, η αλυσίδα διανομής ή ο λιανέμπορος, γιατί δυστυχώς οι τιμές παραγωγού είναι πολύ χαμηλές. Το μεγαλύτερο τμήμα της τελικής τιμής το καρπώνονται οι μεταποιητές και οι ε, διανομής, οι λιανέμποροι. Και αυτοί υπαγορεύουν τους κανόνες. Θέλουμε λοιπόν υποχρεωτική επισήμαση, ώστε εγώ, ο καταναλωτή που θα αγοράζω ένα προϊόν, να ξέρω τι τμήμα τη τιμή πηγαίνει στον παραγωγό, στον Γιώργο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Πάνω από 20 συνάδελφοι έλαβαν το λόγο. Μα, συγγνώμη, πρώτος ήσασταν στον κατάλογο, αλλά παραιτηθήκατε. Α, κατάλαβα καλά, κύριε Ντές. Παρακαλώ. Κύριος Γιάς, ο κύριος Δες, πρόεδρε. Ε, δεν ζήτησα το λόγο πριν, γιατί ήθελα να κάνω κάποια τηλεφωνήματα και ήθελα να ακούσω και τις ομιλίες. Αυτό δεν ήθελα να μιλήσω. 40 χρόνια μιλάμε για τα θέματα της τιμής. Εγώ την γερμανική αγορά τη γνωρίζω πιο καλά βεβαίως. Η κατάσταση για τον παραγωγό επιδεινώνεται διαρκώς από χρόνο σε χρόνο και είναι προφανές ότι δεν μπορεί ο παραγωγός να συμμαχίσει με άλλους παραγωγούς ε, σε τόσο μεγάλο αριθμό και όγκο ώστε να βρίσκεται σε πεδίο ισότιμο με τον ε, Λιανό πολιτή και να μπορεί να διαπραγματεύεται επίσης ώρες. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα, μέτρα σκληρά όπως ε, έχουμε κάνει και στην περίπτωση των ε, τηλεοπικοινωνιών και των ομίλων που επέβαλαν υψηλά τέλη ε, περιαγωγής. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τον ε, γεωργικό τομέα και το διατροφικό τομέα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα όμιλο στην Ευρώπη που να έχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από το 10%. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να ορίσουμε αυστηρούς κανόνες με συγκεκριμένα ποσοστά και θα εξασφαλίσουμε έτσι τις συνθήκες ισότητας αγοράς. Να είναι ξεκάθαρες λοιπόν οι συμβάσεις οι οποίες θα μιλούν και για, τα, ε, για τις ποσότητες που θα παραδίδονται. Εάν έχω ε, συμφωνήσει ε, μία ποσότητα ε, που έχει παραγάγει ο συνεταιρισμό μου ε, και να την παραδώσω στα δε τιμή. Αλλά μετά ε, πέφτουν οι τιμές στην αγορά. Ο αγοραστής, ο ενδιάμεσολαβητής, βρίσκει χίλιες δικαιολογίες για να μην αγοράσει το προϊόν. Ε, λοιπόν πρέπει να πιέσουμε τους μεγάλους ομίλους και εγώ το λέω που είμαι από συντηρητικό κόμμα πως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση και δεν μπορούν να ε, χρησιμοποιούν τις συνθήκες της αγοράς κατά τον τρόπο αυτόν. Τέλειωσα. Ναι, αλλά έτσι πετάτε το μπαλάκι σε μας. Μας ε, ρίχνετε πίσω το μπαλάκι, γιατί πριν από τρία χρόνια το είχαμε προτείνει. Γιατί δεν είχαμε επιχειρήσει τότε πριν από τρία χρόνια να το υιοθετήσουμε. Ε, μοιραστείτε το χρόνο μεταξύ σας. Έχετε 20 λεπτά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία. Είναι μια πλημμυρίδα ερωτήσεων αυτή. Δεν θα απαντήσω πιστεύω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, αν αυτή ήταν η πρόθεση, προφανώς δεν θα είμαι σε θέση. Όμως να τονίσω κάποια από τα στοιχεία που προέκυψαν από την συζήτηση. Πολλοί από τους ερωτώντες τα επεσήμαναν. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της σταθεροποίησης των τιμών και του επίπεδου των τιμών για τη σταθεροποίηση. Μπορεί κανείς να προβλέψει μέσα για να υπάρχει μικρότερη διακύμανση. Όμως τα μέσα αυτά μπορούν σε πολύ μικρό βαθμό να επηρεάσουν το επίπεδο των τιμών. Το επίπεδο των τιμών είναι συνέπεια της παροχής στην αγορά της προσφοράς στην αγορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ουσιαστική διαφορά όταν συζητάμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν θέλει κανείς να ε, κάνει τις τιμές σταθερές, μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Αν όμως θέλει να τις αυξήσει, πρέπει να κάνει πράγματα πιο διαφορετικά, να παρέμβει στην αγορά. Ε, τώρα ας πούμε ότι έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε παρεμβάσεις και λόγω των αλλαγών στην ΚΑΠ έχουμε αλλάξει το σύστημα για να έχουμε όλο και λιγότερες παρεμβάσεις στην αγορά και όλο και λιγότερη παρέμβαση από τα κράτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αγορά, δηλαδή περισσότερη διαχείριση από τις κεντρικές αρχές. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Είναι η βασική διαφορά μεταξύ της σταθεροποίησης των τιμών και της μόρφωσης, ε, της διαμόρφωσης των τιμών, του επίπεδου που φτάνουν. Το δεύτερο πρόβλημα που εφηγεί είχε να κάνει με τον κοινό παρανομαστή των προτύπων. Αυτή είναι σημαντική κέρια παρατήρηση, διότι παράγουμε γάλα, παράγουμε χείριο κρέα. δημητριακά. Ομογενή, α πούμε, αγαθά, τα οποία είναι ανταλλάξω με άλλα προϊόντα από τον κόσμο. Εάν συνεχίσουμε να παράγουμε τέτοιου είδους ομογενή προϊόντα που δεν διακρίνονται λόγω του εμπορικού τους χαρακτήρα, του τοπικού τους χαρακτήρα ή κάποιου άλλου στοιχείου που μπορεί να τα ξεχωρίσει, θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε παντού στον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Άρα ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Εάν όμως θέσουμε πρότυπα, θετικά πρότυπα, πρότυπα προέλευσης ας πούμε, ή ζωικής ευζοίας και το καθεξής και βάλουμε και την ανάλογη σήμανση στα προϊόντα, αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση που έγινε για την ε, αναγκαστική σήμανση, τότε αλλάζουν οι δυνατότητες. Όμως ξέρετε, μιλάμε για την ποιότητα, την ενίσχυση της ποιότητας και το πώς θα διαφύγουμε από το φαύλο κύκλο τη ε, της ομογένειας των προϊόντων. Εδώ και 30 χρόνια το συζητάμε και προσπαθούμε ακόμα και παράγουμε. Παράγουμε ακόμα ομογενή προϊόντα. Νομίζω η βασική υποχρέωση εδώ για τους παραγωγούς είναι να επιλέξουν τι θέλουν. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τις μικρού μεγέθους και μεσαίου μεγέθους και μεγάλες επιχειρήσεις στη Γεωργία. Είναι προφανές ότι τα γενικά μέτρα για να ε, αντιμετωπίσουμε την επίδραση της ε, παγκόσμιας αγοράς είναι κάτι διαφορετικό από το να προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο από τους μικρομεσαίους παραγωγούς στην Ήπεθρο. Είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα αυτά. Γι' αυτό όταν ε, είχα αναλάβει καθήκοντα στις κάτω χώρες, είχα υπερασπιστεί την ιδέα ότι χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τις περιφέρειες που έχουν σημασία για την διατήρηση του τοπίου, για την προστασία της φύσης ή τέλος πάντων που σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες μπορούν να συνεισφέρουν στο γενικό καλό, πέραν των συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων. Αυτό είναι ένα είδος πολιτικής που εδώ στην Ευρώπη έχουμε ακολουθήσει με την ανάπτυξη της πολιτικής της υπαίθρου. Δεν είναι πολύ λογικό να έχουμε ένα είδος πολιτικής, ακριβώς το ίδιο για όλου, όλου το μεγέθος της όλο το μεγεθόν της εκμεταλλεύσης. Οι μεγάλες εταιρείες επικεντρώνονται στην παγκόσμια αγορά και το διεθνή ανταγωνισμό και βεβαίω πρέπει να κάνουν και αυτή τη δουλειά του και αν αυτό θέλουν να κάνουν θα πρέπει να του αφήνουμε. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν κιόλα ότι πρέπει να αναλάβουν το βάρο τη επιλογή του και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τα εργαλεία που συζητήσαμε στην ομάδα δράσης μπορεί να βοηθούν κάποιες εκμεταλλεύσεις. ή μικρότερες σίγουρα ε, χρήζουν διαφορετικών εργαλείων αντιμετώπισης. Και θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους προϊόντα μπορούν να προσφέρουν ε, στο κοινό, στο καταναλωτή. αλλά θέλουμε να εξασφαλίζουν ένα ε, εισόδημα προσφέροντας ακριβώς υπηρεσίες για όλους. Έπειτα, το δίκαιο ανταγωνισμού, τέταρτη παρατήρηση. Αυτό είναι σίγουρα από τα βασικά. Όμως, ε, μία παρατήρηση πρέπει να κάνω ευθύς εξ αρχής, ως Γεωργός, παρόλο που αμφισβητήθηκε αν είμαι πραγματικά Γεωργός, αλλά σας διαβεβαιώ είμαι και να υποφεληθώ για να απαντήσω σε εκείνον που είπε ότι δεν υπάρχει καμία γεωργία, για ελάτε να αρμέξουμε μια γελάδα και θα σας πω ποιος θα τα πάει καλύτερα, ε? Εντάξει, 30 χρόνια αρμέγω. Δεν έχω πιστοποιητικό ίσως, αλλά σας πάω στοίχημα. Δίκαιο ανταγωνισμού. Για το δίκαιο του ανταγωνισμού, σίγουρα είναι ένα θέμα αλλά δείτε το και από την άλλη πλευρά. Πώ μπορούν οι γεωργοί να συνεργάζονται. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Φυσικά έχουμε συνεταιριστικέ οργανώσει, αλλά έχουμε πολλέ. Πώ να του δώσουμε κίνητρα να οργανώνται οργανώνονται περισσότερο σε συνεταιρισμού από ό,τι στο παρελθόν. Ήδη αυτό συμβαίνει σε έναν βαθμό. Γι' αυτό μιλάμε για δίκαιο Πρέπει να ξεκινήσουμε πάντως με την επιθυμία, την προθυμία των γεωργών να δώσουν τα χέρια και να ενωθούν. Να ενωθούν και να δημιουργήσουν σχηματισμούς παραγωγών. Τότε αρχίζουμε να μιλάμε. Και βεβαίω τότε το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι κάτι που μπορεί να αρχίσει να μα απασχολεί. Για αυτού του είδου του συνεταιρισμού, το δίκαιο του ανταγωνισμού θα ισχύει διαφορετικά σε σχέση με τι μεγάλε εταιρείε. Σίγουρα είναι ένα ζήτημα, ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά μην ξεκινάμε από τη λάθος άκρη του όλου ζητήματο. Σα διαβεβαιώ ότι όλε τι παρατηρήσει που κάνατε τι έχω λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Ένα στοιχείο για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Η εισηγήτρια, κυρία Μαγκίνες το είπε, και θα ήθελα να το σχολιάσω κι αυτό, αλλά κάπως λεπτομερέστερα με την ίδια και επειδή ένα σχετικό ερώτημα έθεσε και ο κύριος Νταντέν. Ίσως ε, να έχουμε την ευκαιρία σε μια πιο σύντομη συζήτηση μεταξύ μας για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Θα ήταν καλή ιδέα, πιστεύω. Και μερικές τελευταίες απαντήσεις από πλευρά μου, μετά θα στραφώ στους συναδέλφους για ενισχύσεις. Ε, η τελευταία παρατήρηση του κυρίου Ντες ο οποίος με τέτοια εφράδια και πυγμή μίλησε για το τι θα πρέπει να γίνει. Ναι, η παραγωγή είναι σίγουρα πιο αδύναμη και σίγουρα δεν έχουν ενισχύσει τη θέση τους. Όμως, όπως είπα προηγουμένως, οι ίδιοι παραγωγοί έχουν στα χέρια τους την επιλογή να σταθούν και ε, στο ύψος τους και να έχουν περισσότερη συνεργασία μεταξύ τους. Έπειτα μιλήσαμε για τις απογοητεύσεις που προκαλεί το δίκαιο προς ο πρόσκομα για να επηρεάσουμε καλύτερα τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω βέβαια σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Τις έχω όμως σημειώσει και θα τις εξετάσω όσο προχωράνε οι συζητήσεις. Γιατί πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερο τη ε, συμβολή των μελών του Κοινοβουλίου και της δική σας Επιτροπής όλο ιδιαίτερος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε ε, ε Χόισλινγκ, δέχεστε την πρόκληση για να πάτε να αρμέξετε γελάδες. Äh, Πρόεδρε, ευχαρίστω. Και εγώ έχω μια γελαβίτσα δικιά μου. Το αποτέλεσμα όμως τι θα είναι, αυτό είναι το ερώτημα. Τι κρίνεται δηλαδή. Παρακαλώ. Κύριος Μπιτζή. Ευχαριστώ. Α, θα μιλήσω γαλλικά, αν μου το επιτρέπετε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης και για την ευκαιρία που μας δώσατε να ανταλλάξουμε απόψεις. Βέβαια, ο καθένα διορίστηκε προσωπικά σε αυτή την ομάδα εργασία. Εγώ εκπροσωπώ βέβαια τις επιχειρήσεις ε, ανάμεσα, που ήταν ο, ο στόχος πολλών σχολείων. Ε, και πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Το αντανακλαστικό που έχουμε μερικές φορές ε, και αυτό το νόημα είχαν και πολλά σχόλια και είπαμε καλό που γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ο αυτοματισμός λοιπόν που έχουμε μερικές φορές είναι ότι ε, ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα ε, καταπληκτικό δυναμικό αγροεπιστηστικής παραγωγής. Έχουμε ένα φάσμα παραγωγών, τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων, Έχουμε τοπικές σπεσιαλιτέ, και πολύ εκλεπτισμένα προϊόντα σε πολλούς τομείς παραγωγής και αυτό που διαπιστώνουμε στα καταστήματά μας και παντού είναι ότι όσο καλά πάντα πράγματα, τόσο οι καταναλωτές απαιτούν ποιοτικά, τοπικά προϊόντα και γι' αυτό χρειάζεται ειλικρινής ε, και αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό το σημείο είναι θεμελιώδες. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τους μηχανισμούς που ενισχύουν την προστιθέμενη αξία των αγροεπιστηστικών προϊόντων. Πριν από λίγο αναφέρθηκε ο Ίνος και οι τομείς που ακολούθησαν τέτοιες στρατηγικές είναι αυτές που λειτουργούν καλύτερα και που ξεπερνούν πιο εύκολα τις κρίσεις από άλλους τομείς. Αυτό είναι το πρώτο μου σημείο, το πρώτο σημαντικό σχόλιο. Το δεύτερο είναι, που είναι σημαντικό είναι ότι τα γεωργικά προϊόντα δεν μπορούν να τύχουν ε, τις ίδιες διαχείριση με οποιαδήποτε άλλο τυχαίο προϊόν. Τα μέτρα προσαρμογή είναι πολύ πιο δύσκολα να εφαρμοστούν για τις γεωργικές παραγωγές και κυρίω ε, για τα προϊόντα τη κτηνοτροφία. Ε, και η κτηνοτροφία είναι ο κλάδο που καταξοχήν αντιμετωπίζει την κρίση. Και ο κτηνοτρόφος τα βρίσκει πολύ σκούρα γιατί πρέπει να μειώσει το ζωικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να προσβέσει τις επενδύσεις του. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των γεωργικών προϊόντων. Και επίση, ε, οι διακοιμάνσεις που υφίστανται σε διεθνές επίπεδο, οι περιβαλλοντικές διακοιμάνσεις είναι τεράστιες. Τώρα δεν έχουμε άποψη για το ποιε είναι οι καλύτερε αγορέ για να ορίσουν τι τιμέ. Θεωρούμε όμω ότι θα πρέπει συλλογικά να υπάρχει δυνατότητα διαχείριση ε, τη σπανιότητα των προϊόντων. Δηλαδή, να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο παρακολούθηση τη προσφορά των προϊόντων στην αγορά, γιατί οι τιμέ είναι χαμηλέ όταν υπάρχουν ανισορροπίε στην αγορά μεταξύ προσφορά και ζήτηση. Και όταν είναι υψηλέ τιμέ των σιτηρών ή όταν η τιμή του γάλακτο ε, είναι υψηλή γιατί οι βιομηχανικές τιμές είναι καλές και αυτούν και οι εξαγωγέ. Πολλοί λένε χάρη στα μεγάλα σούπερ μάρκετ είναι υψηλέ οι τιμέ. Όταν είναι όμω χαμηλέ οι τιμέ, τότε λένε αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ για αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει όμω να βρούμε μια ισορροπία. Μια ελάχιστη ισορροπία στι αγορέ. Και από αυτήν την άποψη η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική ε, το παρατράβηξε και δεν επέτρεψε την δημιουργία ενό τέτοιου μηχανισμού. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε επισταμμένος στην ομάδα μας, στην ομάδα εργασίας μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τρίτο στοιχείο, κατά τη γνώμη μου χρήσιμο, είναι το πώς θα λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες, επιχειρηματικές ανάγκες των γεωργικών ε, επιχειρήσεων, γιατί Τη σήμερα ημέρα ε, συνυπάρχουν οι μικρέ και οι μεγάλες επιχειρήσεις και μπορεί οι μεγάλες επιχειρήσεις να φαίνονται πιο ρωμαλές και στιβαρές αλλά μπορεί αυτό να είναι ένα απλώς φαινόμενο ε, να μην ισχύει στην πράξη. Θα πρέπει να μπορούν όλε οι επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά του Αν δούμε τα προβλήματα τη κτηνοτροφίας, της γαλλικής κτηνοτροφίας. Βέβαια, η Καρφόρ έχει καταστήματα σε έξι χώρε μέλη και έχουμε επαφές στις χώρες αυτές, αλλά σε πολλές ε, χώρες τα προβλήματα της επιχείρησης δεν ε, έχουν λυθεί. Και είναι σίγουρος ο δρόμος προς τη δυσκολία και την αντικσότητα. Δεν μπορούμε με υψηλά χρέη να τα βγάλουμε πέρα. Και διαπιστώνουμε σήμερα ότι πολλές επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες και το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Επίσης, ε, έχουμε στις επιχειρήσεις κάποια συστήματα μείωσης κινδύνου με τις ασφαλίσεις ε, ή συστήματα εγγύσεων. Περνάμε πολύ χρόνο στην ανάλυση των κινδύνων και στην αναζήτηση μέσων και μηχανισμών για να περιορίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί η επιχείρηση είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να τους προλαμβάνει να τους αποτρέπει να τους αποσοβεί όταν ε, παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Οπότε έτσι θα λάβουμε ταυτόχρονα υπόψη και μερικές από τις ανησυχίες των Γιώργων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγούσον, χαίρομαι που είμαι εδώ, πρώτη φορά μου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με το δικό μου τομέα δραστηριοποίησης της προθεσμιακής αγοράς και τα παραγωγά. Και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ωφελήσει τον ε, μικρό παραγωγό ή αν είναι λύσεις διαχειριστικέ μόνο για τους μεγαλύτερου παραγωγούς ε, οι προθεσμιακές αγορές να σα πω, οι μεγαλύτεροι αξιοποιούν τι προθεσμιακέ αγορέ, οι δε μικρότεροι μέσα από του συνεταιρισμού του ή κάποιε άλλε επιχειρησιακέ συμβάσει, ε, ενοποιούν τι δυνάμει του και επιλέγουν είτε να πωλήσουν μέσα από ένα συμβόλαιο ε, ε, προθεσμιακό που κοιτάει δηλαδή προ το μέλλον είτε κατά περίπτωση. Το προθεσμιακό εξαρτάται βέβαια από τι προθεσμιακέ αγορέ, εφόσον βέβαια βρίσκουν την κατάλληλη αγορά. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή πιο χρήσιμες για τον μικρότερο παραγωγό. Για κάποιους βέβαια δεν είναι δυνατόν να αξιοποιήσει καθόλου τις προθεσμιακές αγορές. Και μια και έγινε τόσο λόγος για το γάλα. Στη Σουηδία έχουμε μια μεγάλη γαλακτοκομική εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια, πολύ αποτελεσματική, και πάει σε αυτήν όλο το γάλα και κάνει πολύ καλό γάλα. Αν ας πούμε οι Γάλλοι, οι Ιταλοί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο με το κρασί τους ή και οι άλλοι που παράγουν δεχμένο κρασί, δεν θα ήταν καλύτερα. δεν θα μπορούσε ένας μικρός παραγωγός ε, να χρησιμοποιεί προθεσμιακές αγορές για χίδιν σαρτονέ. Ίσως όχι. Η άμεση, η άμεση κρίση τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις χαμηλές, με τις χαμηλές τιμές. Καθήκον μας είναι να κάνουμε κάποιες προτάσεις πολιτικής που θα χρειαστούν χρόνο. Και άρα δεν να έχουν στόχο να καλύψουν την τωρινή κρίση. Διορθώστε μου αν Οι προθεσμιακές αγορές σαν στόχο έχουν και να αποτρέψουν τον κίνδυνο, να μετακυλήσουμε τον κίνδυνο του παραγωγού σε κάποιον άλλον. Κάτι αντίστοιχο με την ενέργεια είναι αυτός ο κίνδυνο. δηλαδή μετατρέπεται, κινείται, αλλά δεν εξαντλείται, δεν χάνεται. Ε, εάν δηλαδή δεν την ε, μεταφέρει κάπου, ε, δεν τον μεταφέρει κάπου κίνδυνο ο παραγωγός, θα μείνει σε αυτόν. Κοιτάει λοιπόν προς τα μπρος και ορίζει μια τιμή για το μέλλον, ένα τρόπο εξορρόπησης, αλλά και ε, διάθεσης πλεονασματικών αποθεμάτων. Είναι καινούρια αυτή η αγορά για τα γαλακτοκομικά. Το 2011 μόλις ξεκίνησε. Χρειάζεται βέβαια κάποιο χρόνο ρονταρίσματος. Ο βουλευτής του Ρωμαίου Βασιλού νομίζω έχει φύγει, αναφέρθηκε στο ΜΕΦΙΤ 2. Την οδηγία. Και άλλη δουλειά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα επηρεάσει αυτή την κατάσταση. Αυτά νομίζω είχα να πω εγώ από το τομέα μου. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι, ότι αξίζει να εξετάσουμε την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά και πώς επηρεάζεται από τους εξωτερικούς παράγοντες, γιατί δεν είμαστε απομονωμένοι, εξαρτώμαστε από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Αν αγνοήσουμε αυτές τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που διαμορφώνονται σήμερα μέσω ε, παγκόσμιων συμφωνιών, TTIP, Mercosur, ΣΥΤΑ, με τον Καναδά, Συμφωνία Εμπορική με τη Νέα Ζηλανδία. Αν δεν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, τότε χαίρεται ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Ή λοιπόν ε, ε, θα υιοθετήσουμε απόλυτα φιλελεύθερες αρχές και προδιαγραφές εμπορίου, δηλαδή όλα ανοιχτά, ανοιχτές αγορές, ή θα περιχαρακώσουμε κάπως ε, και θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Επίσης, ε, η κατακόρυφη ολοκλήρωση. Νομίζω ότι μεταξύ άλλων μία από τις επιτυχίες ε, του σχετικού μοντέλου είναι αυτή η κατακόρυφη ολοκλήρωση. Η κατακόρυφη ολοκλήρωση όμως πρέπει να προσδιορίζει το, ξεκάθαρα το ρόλο μεταξύ του παραγωγού, του μεταποιητή και του εμπόρου και γι' αυτό χρειάζονται κανόνε. Θα πρέπει να θεσπιστούν αυτοί οι κανόνε. Αν οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, οι χρηματοοικονομικέ αγορέ δεν είναι σε θέση να ε, βάλουν μια τάξη σε αυτό το σύστημα και γίνει, ε, ε, φτάσουμε σε μια κρίση. Φανταστείτε, φτάσαμε κρίση στον τραπεζικό τομέα που ήταν πολύ πιο εύκολη η ρύθμιση, πόσο πιο δύσκολη είναι η ρύθμιση στο γερικό τομέα που εξαρτάται και από το περιβάλλον και εκεί οι διακοιμάνσεις είναι πολύ πιο απότομες. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγισης μας, τη σκοπιά μας, την τον τρόπο σκέψης μας και να ευθύσουμε μια νέα θεώρηση για τα θέματα αυτά. Περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς το πόρισμα της ομάδας εργασίας σας και τα αποτελέσματα του έργου σας. Επίσης περιμένουμε τα πορίσματα και του υψηλού ε, φόρουμ για τα θέματα αυτά και ελπίζω να έχετε κάποια συνάφεια στις εργασίες. Πάντως ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση, διατυπώθηκε πληθώρα ερωτήσεων και θα ήθελα να παρακαλούσα τους συναδέλφους να στείλουν και γραπτό στις ερωτήσεις τους μέσω της γραμματείας στην ομάδα εργασίας του κ. Βέρμαν. Νομίζω έτσι θα βοηθείτε και εσείς να σας στείλουμε ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Μας αναγγείλατε για το φθινόπωρο την έκθεσή σας. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη λοιπόν αυτή η ανταλλαγή απόψεων, γιατί το θέμα είναι πολύ δύσκολο. αλλά ταυτόχρονα είναι και υψηλέ οι προσδοκίε. Και αυτό είναι ο ρόλο τη Επιτροπή μα, να ασχολείται με δύσκολα ζητήματα. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρατηρήσει ή ερωτήσει, να ευχαριστήσω και πάλι θερμά του καλεσμένου μα, του εμπειρογνώμονε. για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σε αυτό το ιδιαίτερο δύσκολο ζήτημα. Θα ήθελα, πριν ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη, να εγκρίνουμε ε, τα πρακτικά και τις αποφάσεις των συντονιστών από την προηγούμενη συνεδρίαση. Τη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθώ ότι εγκρίνονται. Στα διάφορα Θα ήθελα να ζητήσω από τους Ολλανδούς συναδέρφους να κάνουν ένα διάβημα προς την Ολλανδική Προεδρία για το θέμα της αμμονίας, γιατί οι εξελίξεις δεν είναι καθόλου ε, θετικές. Η Προεδρία θέλει να ε, κάνει πιο αυστηρές προδιαγραφές. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το θέμα. Η επόμενη συνεδρία 24 Μαΐου. Κυρία Αγγιλέρα, ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ στη συνεδρίαση των συντονιστών. Εδώ το βλέπω, αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει όταν το συζητούσαμε, ότι εγκρίναμε την προφορική ερώτηση μετασυζητήσεως. Δεν είχα καταλάβει ότι, θα, ότι εγκρίναμε αυτή την προφορική ερώτηση. Αν οι άλλοι την κατάλαβαν με αυτό το περιεχόμενο, τώρα, τότε μάλλον εγώ κάνω λάθος. Τώρα βλέπω όμως την τελική διατύπωση και εγώ ομολογώ ότι δεν είχα καταλάβει ότι αυτό θα ήταν το περιεχόμενο. Δεν είχα καταλάβει λοιπόν καλά την πρόταση για προφορική ερώτηση με συζήτηση. Ποια προφορική ερώτηση λέτε? Έχουμε στα πρακτικά στις αποφάσει των συντονιστών μια προφορική ερώτηση για την ύπαρξη μη δασμολογικών φραγμών στην εσωτερική αγορά. Αυτή η προφορική ερώτηση ήδη είχε γίνει. Δεν είχε μπει στην Ολομένη και τώρα την ε, συμπεριλάβαμε στα πρακτικά ως απόφαση των συντονιστών. Δεν το είχαμε πει ρητά. Θα ήθελα να το διευκρινίσω γιατί εγώ άλλα είχα καταλάβει. Τι γίνεται με την ερώτηση. Πώς το είχαν καταλάβει οι συντονιστές. Εγώ είχα πει ότι είχε υποβληθεί ως προφορική ερώτηση. Αυτή είναι δική μου πρόταση. Να υποβληθεί ως προφορική ερώτηση. Αλλά είμαι ανοιχτό σε συζήτηση αν θα πρέπει να το θέσουμε ή τι περιεχόμενο να δώσουμε. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι μας κάλεσε στις 6 και 4 στον τρίτο όροφο μπροστά στο εστιατόριο στις 6 και 4 για μια σεμνή δεξίωση. Στο ίδιο κτίριο, στον τρίτο όροφο. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, ραντεβού στις 24 Μαΐου για την επόμενη συνεδρίαση. Και εκεί θα μιλήσουμε για την αγορά του γάλακτος. Είναι αρκετά πλήρες το πρόγραμμα και τις επόμενες συνεδρίασεις. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονε, σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας απόγευμα.